Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε, να συμμαζευτούμε λίγο, λέει ο Πρόεδρος. We are up to item six on the... Έχουμε φτάσει στο σημείο 6 της ε, ημερησίας διάταξης και αναφέρεται στον ορισμό εισηγητών. Πρώτη ανακοίνωση είναι ότι όσοι συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία που θα πάει αύριο στην Αυστρία, στη Σλοβενία και την Κροατία, να πω ότι αναμένεται μία απόφαση. Ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία προειδοποίηση των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας ότι ε, θα ε, ξεκινήσουν απεργία. Επομένως, ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα αύριο να φύγουμε από τις Βρυξέλλες. Θα σας κρατήσω ενήμερους βέβαια. αλλά εάν πραγματοποιηθεί η απεργία δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε. Ε, θα σας έχω την απαραίτητη ενημέρωση ο κύριος Αϊδελ Κατράουι προσπαθεί να πιέσει με όλη του τη δύναμη έτσι ώστε και με όλη την επιρροή που διαθέτει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ε, ε, επίσκεψή μας. Αλλά ε, τι να σας πω, εάν πραγματοποιηθεί η απεργία των ελεγκτών τότε δυστυχώς τι να κάνουμε. Να αναφερθώ τώρα στην συνεδρίαση των συντονιστών. Πρώτα απ' όλα ο ορισμός εισηγητών και ε, λοιπόν εισηγητών είναι απόφαση λοιπόν των, ε, το, των συντονιστών όσον αφορά τους ε, σιδηροδρόμους να το κάνουν οι ε, σοσιαλιστές. Όσον αφορά την θαλάσσια γνώμη 2020, η απόφαση των συντονιστών ήταν να μην συνταχθεί ε, γνωμοδότηση. Θα δούμε τι θα κάνει με την, ε, η, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, με την έκθεσή της και θα δούμε μετά. Όσον αφορά τις επισκέψεις αντιπροσωπιών και τις ακροάσεις, Γίνεται μια πρόταση βέβαια όσο γίνεται να είμαστε πιο κοντά στη, στα συνδικάτα, αλλά, αλλά εν πάση περιπτώσει αποφασίστηκε να επισκεφθούμε την ευρωπεριοχή μας για να δούμε πώς έχουν οι μεταφορές εκεί και γενικά να δούμε πώς ε, ε, είναι οι μεταφορές στον Πενελούξο. Είναι πρόταση των Πρασίνων και του ΕΛΚ. Κοινή πρόταση. Δεύτερη επίσκεψη στο Μαρόκο, πρόταση των σοσιαλιστών. Και εκεί να δούμε τις ε, συμφωνίες ε, μεταφορών μεταξύ ε, Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα την κατάσταση όσον αφορά το δίκτυό τους κτλ. Και ενδεχομένως θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε και τον νέο σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Ραμπάτ με την Ταγκέρη υψηλού uh, μεγάλης ταχύτητας. Και η τρίτη πρόταση είναι μια ας πούμε κοινή πρόταση δύο πολιτικών ομάδων που αφορά μια κοινή ε, μια ε, επίσκεψη ε, και στην γαλλική πλευρά, Λαγκεντό Κρουσιγιόν και στην ισπανική πλευρά μέχρι τη Βαρκελόνη υπάρχουν εκεί προβλήματα όσον αφορά τις μεταφορές, το πέρασμα των συνόρων κτλ. Το, η ομάδα Άλντι έχει, φιλελεύθεροι έχουν προτείνει την επίσκεψη αυτή. Αυτά όσον αφορά το 2011. μετά από πολλή συζήτηση όσον αφορά το κατά πόσον οι ακροάσεις αξίζει τον κόπο να οργανώνονται, τρεις ε, ομάδες υπέβαλαν αρκετές προτάσεις. Και θα υπάρξουν τρεις προτάσεις λοιπόν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα έτσι ώστε να γίνει σεβαστή και η χρονική προθεσμία που υπάρχει. Τρεις ήταν οι ομάδες, το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές και το ΑΛΔΕ που έκαναν κάποιες ε, προτάσεις. Θα εκπονηθεί λοιπόν ένας κατάλογος, ο οποίος θα αποτελέσει και τη βάση για τις ακροάσεις που θα οργανωθούν το 2011. Βεβαίως ε, ε, μπορούμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε, να διαφοροποιήσουμε. Απλώς θα αποτελέσει μια πρώτη βάση. Όσον αφορά την επιτροπολογία, Ο κύριος Αλκαντράουι, ένας από τους ε, εισηγητές μας, ε, μας ε, κοινοποίησε, μας ενημέρωσε για δύο TSI για, την, για τους σιδηροδρόμους και ενδεχομένως να υπάρξει αυτή η συζήτηση σχετικά με να είναι ένα βήμα παρά την ενιαία ε, τιμολόγηση και ε, έκδοση εισιτηρίων, σύστημα δηλαδή έκδοση εισιτηρίων. Ε, όταν ολοκληρωθούν οι προτάσεις τον Οκτώβριο θα υποβληθούν στην Επιτροπολογία πριν φτάσουν στο Κοινοβούλιο. Συμφωνήθηκε από τους συντονιστές επίσης ότι ε, θα οργανωθεί και μία ακρόαση για την εφαρμογή GNSS κάποια στιγμή. Ενδεχομένως ε, προς τα τέλη του Νοεμβρίου, σε δύο μήνες δηλαδή, να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης, συζητήσεις ε, για την κρίση και για την ε, φτώχεια 18-19 Νοεμβρίου ε, ζητήθηκε να εκπονηθεί ένα έγγραφο για την ε, αγορά και για τους τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης και της φτώχειας. Υπάρχει και εδώ χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου και επομένως θα πρέπει να υποβληθεί το έγγραφο αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του μήνα. Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το 2011 το έχετε στο φάκελό σας, φαντάζομαι το έχετε ε, συμβουλευθεί. Υπό τα διάφορα ε, υπήρξε ε, μια πολύ σημαντική συζήτηση για το όριο του 0,1 στη Βαλτική θάλασσα που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Θαλάσσια Ομοσπονδία και δόθηκαν πληροφορίες ε, σχετικά ε, με το θέμα αυτό. Ε, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης επιπτώσεων και όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ξανά το θέμα. Συζητήσαμε και το θέμα της Προεδρίας της IB και επίσης συζητήσαμε και για το θέμα της ανταλλαγής ε, επιστολών ε, με θέμα την απελευθέρωση των ε, ουρανών, επιστολές που είχαμε, που ανταλλάξαμε και με, τον, με την Επιτροπή Ελευθεριών. Η Κεντρική Επιτροπή Πλεύσης του Ρήνου ζήτησε μια συνάντηση ε, μαζί μας ε, στη διάρκεια της ε, Ολομελίας του Στρασβούργου τον μήνα Ιανουάριο, 19 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνάντηση. ο αντιπρόεδρος Βαντάλ αρχικά είχε κάνει την πρόταση, δηλαδή να επισκεφθούμε τον Ρήνο και τα γραφεία της Ένωσης αυτής. Επίσης, όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση ε, σχεδίων και προγραμμάτων για τις μεταφορές και όσον αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ε, επιβατών στον τομέα των σιδηροδρόμων. Ε, είχαμε ανακοινώσει τη Επιτροπή από αυτόν και θα στείλω επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο Κάλλα για να δω ακριβώς περί τίνο πρόκειται. Τέλος, ε, σε συνέχεια της προφορικής ερώτησης ε, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η πλειοψηφία λέει ότι δεν θα υπάρξει, δεν θέλει να υπάρξει συνέχεια και επομένως η πρόταση καταψηφίστηκε. Αυτά ήταν ε, που είχα να σας πω σχετικά με την αναφορά ε, που ήθελα να σας κάνω για την ε, συνάντηση των συντονιστών. Δεν βλέπω να έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις από αυτών που μόλις ακούσατε, επομένως άψογα μπορούμε να συνεχίσουμε. Κουράστηκα ήδη, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενο, σημείο στην σε διάταξη. <coughs> Ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία για την ολοκληρωμένη πολιτική θάλασσας. Έκθεση Μάισνερ. Είστε έτοιμοι για να ψηφίσουμε. Έχετε όλοι μαζί τις κάρτες σας. Θα κάνουμε έναν έλεγχο πρώτα. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Είναι καταπληκτικός ο Μπράιαν Σίμψον η ερώτηση για τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Βλέπω 77 κατά. Βλέπω την κυρία Φώστερ να σπέβδει να τροποποιεί την ψήφα της. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ του εαυτού μου. Φαντάζομαι θα έχω μόνο μία ψήφο υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Α, εντάξει, είμαι πιο δημοφιλής από ό,τι φανταζόμουν. Εντάξει, γραμματεία, ως προς την εκπροσώπηση. Αρχίζουμε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι για την τροπολογία 98 έχει αποσυρθεί, γιατί έχει συγχωνευτεί με την 97. Ωραία, η 98 αποσύρεται. Την έχω στην 7η σελίδα του καταλόγου. Για την παράγραφο 29β, έτσι. Όχι, η 98 συγχωνεύεται με την 97 ουσιαστικά. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ναι, ναι, ναι, αλλά σε ποια παράγραφο αναφέρεται. Στην 29β αναφέρεται η τροπολογία 98, για να ξέρουν τα μέλη τι ψηφίζουν. Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαέξι. Προφορική τροπολογία της ηγήτριας. Περιλαμβάνεται στο κατάλογο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Grandes Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχο για τη 19. Άρχεται η ψηφοφορία. As everybody voted, vote is closed. Ψηφίσατε όλοι. τέλο ψηφοφορία. 26 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Είναι αρκετά περίπλοκη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 του κυρίου Τέιλορ. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Για να περιλάβει το, την επιλογή μέχρι το directive ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα μέχρι γεωτρήσεις ε, σε μεγάλο βάθος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, να περιλάβει ε, εκμετάλλευση και τα λοιπά μέχρι την οδηγία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26, Φλέκενστάιν. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 21 ψήφισαν υπέρ και 18 κατά. Εγκρίνεται. 28, Τέιλορ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 φύς. Πες, συγγνώμη. Πε, της Επιτροπής Ελίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί το ΕΛΚ δεν ψήφισε ενωμένα. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 16 της Επιτροπής Αλίας. Τέλος. Δίκιο είχατε. 19 ψήφισαν υπέρ και 20 κατά, άρα απορρίπτεται. 29. Σε τμήματα, δύο τμήματα. Και υπάρχει και προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Δεύτερο τμήμα δηλαδή που αφορά το τρίτο εδάφιο μάλλον. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα που αφορά το τρίτο εδάφιο. Άρχεται η ψηφοφορία. As everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Με ισοπαλία 19. Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε τώρα στην τρίτη συμβαστική τροπολογία κατευθείαν. We now have to vote on the third part, which is support the port infrastructure. Για την υποστήριξη ανάπτυξη των λιμένων. Τρίτο τμήμα στην 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία σε γάμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκα, τροπολογία 18, Αλία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Με την προφορική τροπολογία της ηγήτρης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περιφερειακή Επιτροπή. Δύο τμήματα μέχρι τις ειδικές λύσεις. Το πρώτο τμήμα της πέμπτης τροπολογίας. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα έχει νόημα να το ψηφίσουμε ναι ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 με την προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 της Ελίας ως προσθήκη στην παράγραφο 11. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 43 ως προσθήκη άρχιτη ψηφοφορία ψηφίσετε όλοι τέλος 19 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται 17 της Ελίας ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 Τέιλορ, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν θα ψηφίσουμε την 7. 45 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Πρωτοβουλίες και στρατηγικές στα 47 έχει αποσυρθεί. 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 με την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δύο τμήματα μέχρι τις αυτόνομες περιοχές το πρώτο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, αν έχει νόημα, ναι, υπέρ, κατά, απόχες, Εγκρίνεται. 52 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 με προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 έχει καταπέσει με την πρώτη συμβαστική τροπολογία. 59. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 51. 59, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted, Ψηφίσατε όλοι. Ισοψηφία καταπίπτει, χωρίς αποχές. 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 αποσύρεται. 64 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 αλία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μάλλον έχει εγκριθεί αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 13 της Επιτροπής Αλίας άρχιτη ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος 27 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται. Επόμενο κεφάλαιο, επιτήρηση των θαλασσών. 66 έχει αποσυρθεί, 67 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 αλία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία δέλτα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 78 με την πληροφορική τροπολογία την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι τέλος. 15 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 79 έχει αποσυρθεί, 80. Ποιο Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 σε δύο τμήματα της Επιτροπής Αλίας. Το πρώτο τμήμα μέχρι την προσέγγιση που στηρίζεται στα οικοσυστήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 αποσύρεται. 83 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 83 με την προφορική τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Ε, απορρίπτεται 16 υπέρ, 24 κατά. 85 του κυρίου Τέιλορ με ψηφοφορία κατά τμήματα, δύο τμήματα μέχρι μπορεί εκπομπών. Ποιος είναι υπέρ το πρώτο τμήματος. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Τέλος. Ισοπαλία απορρίπτεται με 20 ψήφους. 84 αποσύρεται, 86 καταπίπτει, γιατί ψηφίσαμε υπέρ του πρώτου τμήματος του 85. Οπότε πάμε συμβαστική τροπολογία ε για την παραγραφή 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί βέβαια τα αρχίζουν και κουράζονται τα χέρια, άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία ε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 27 υπέρ, 13 κατά. Έγκρινεται. Γυρίζουμε σελίδα. Ο πρόεδρος γυρίζει 93. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F, σιγματά. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99, ε, μάλλον 97, 97. Με προφορική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 98 αποσύρεται, 99 ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Η 100 έχει αποσυρθεί, 15 της ε, αλίας σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα μέχρι το υπαρκέστερη χρηματοδότηση, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχέ, απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα, αν έχει νόημα ακόμη, ναι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 101. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 10 άρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Υπέρ 14, 25 κατά. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μια στιγμή τώρα να δούμε τις αλίας 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Πάντα των της υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Πάντα στα ψάρια, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Ευτυχώς λοιπόν για αυτούς που η 12 εμπίπτει στην, στο άρθρο 50, άρα την ψηφίζετε. Πάμε τώρα στην περιφερειακή. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίσως να επαληθεύσουμε γιατί βλέπω ότι το ΕΛΚ δεν ψηφίζει. Ρέτζι 2 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας. Υπέρ 29 κατά 11. Ρέτζι 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 4 όχι λοιπόν τέλος πάντων θα τα πάμε σιγά σιγά 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6, 7, 6 υπέρ συγγνώμη κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ε, επαληθεύσουμε. Ρέτζι 7. Πέρας. 27 υπέρ 14 κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Ωραία. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. 33 υπέρ, 5 κατά και 3 αποχές συγχαρητήρια στην κυρία Μάισνερ. just a minute... Πέντε μόνο λεπτά διάλειμμα. Μετά θα έρθει ο κύριος Γιάννης Όσοι τον γνωρίζετε, θα γνωρίζετε ότι ακριβώς σε πέντε λεπτά θα αρχίσουμε. Colleagues. Φίλες και φίλοι, ας επαναλάβουμε παρακαλώ την συνεδρίαση, προχωρώντας στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, που είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός εναέριος χώρος και με, να ανταλλάξουμε απόψεις με αυτόν τον υπέροχο συντονιστή, που πάντοτε τον θεωρούσα εγώ υπέροχο, αλλά με μεγάλη μου πάντως χαρά τον καλωσορίζω ως πρώην συνάδελφό μας και πρώην αντίπαλο, αλλά πάντως καλό μου φίλο, Τζόρτζ Γιαζεμπόσκι, εδώ στην Επιτροπή μας, στον ρόλο του συντονιστού των λειτουργικών τμήματων του εναερίου χώρου. Έχουμε μέχρι τις 11.30 περιθώριο και είμαι βέβαιος ότι θα εξελιχθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλώς ήρθες, Τζορτζ. Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε και σου δίνουμε αμέσω το λόγο. Στα αγγλικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, είναι πράγματι μεγάλη ευχαρίστηση και για μένα που βρίσκομαι εδώ πάλι. 18 χρόνια πέρασα. Μα είχαμε φτιάξει και τόσα ωραία πακέτα, τον ναυτιλιακό, των σιδηροδρόμων. Είμαστε λοιπόν κάτι σαν ένα είδο εταιρεία πακέτων. Ερχόμαστε τώρα στα ενέργεια είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που υποστηρίξατε τον διορισμό μου, γιατί αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό, διότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είναι φυσικοί σύμμαχοι και το ίδιο φυσικό σύμμαχό σας είμαι και εγώ. Ε, βέβαια πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω την υποστήριξή σας. Διορίστηκα στις 12.08 και περίμενα πάντα με ανυπομονησία αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχει και ένα έγγραφο που ελπίζω ότι σας έχει μοιραστεί, θα σας το εξηγήσω λίγο αργότερα. Ας θυμηθούμε ξανά ποιο είναι το καθήκον, ποια είναι τα καθήκοντα του συντονιστού. Πρώτα να δημιουργήσει αυτά, αυτούς τους ε, τα λειτουργικά τμήματα. Πρώτο λοιπόν. Αλλά μετά από αίτηση των ε, χωρών μελών υποτίθεται να λαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητού μεταξύ των χωρών μελών, εάν υπάρχουν διαφορές. Και τρίτο, θα πρέπει να αναφέρετε σε εσά ένα τρίμηνο. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να με βλέπετε βέβαια κάθε τρίμηνο. Και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται αυτή ε, να αναφέρομαι σε εσά δηλαδή, ως όπλο για να διασφαλίζεται η εφαρμογή των όσων αποφασίζεται. Κάναμε το πρώτο πακέτο, το δεύτερο και τώρα οι χώρε μέλη είναι υποχρεωμένες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσει τους. Εγώ θα παρακολουθώ και θα συμβάλλω στην επίτευξη του στόχου αυτού. Και αυτά τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου, σύμφωνα με τον κανονισμό, τον δικό σας και του Συμβουλίου, έχει χρονοδιάγραμμα. Υποτίθεται ότι αυτά τα τμήματα θα είναι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 έτοιμα. Φαίνεται να είναι πολύ, αλλά δύο χρόνια στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα για την οργάνωση των ε, λειτουργικών τμήματων εναεριού χώρου. Θα θυμάστε στην κρίση που πέρασε το Συμβούλιο, είχε αποφασίσει ότι θα επιταχύνει την διαδικασία δημιουργίας των τμήματων εναερίου χώρου. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό καθήκον και θα εκόμιζα γλάφκα εις Αθήνας αν έπρεπε να εξηγήσω σε εσά περί τίνο πρόκειται. Αλλά τέλο πάντων για τα νέα μέλη α εξηγήσω. Ποιο είναι ο στόχο των ε, λειτουργικών τμήματων ενεργού χώρου. Δεν είναι καθεαυτόν η δημιουργία τους, αλλά έχει τέσσερι στόχους. Πρώτο, βελτίωση τη ασφάλεια στου εθέρε. Δεύτερο, βελτίωση τη χωρητικότητα των εθέρων. Τρίτο, καλύτερη αποδοτικότητα των ε, συστημάτων ενέργειου ελέγχου. Και τέταρτο, οικολογικός χαρακτήρας, δηλαδή φιλικότερος προς το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τις κοινωνικές, την κοινωνική κατάσταση των ε, ε, κοινωνικών εταίρων, των ελεγκτών εν τέλει. Αυτή είναι η στόχη που προσπαθούμε να επιτύχουμε δημιουργώντας τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου είχαμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, τότε με το πρώτο πακέτο, το δεύτερο πακέτο, αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτά τα λεγόμενα με την αγγλική συντομογραφία FAB και είπαμε ότι θα αρχίσουμε ανάποδα. Ως χώρες μέλη που έχουν βεβαίως κυριαρχία στους εθέρες, θέλουμε να το κάνουμε. Έτσι είπαν οι χώρες μέλη. Άρα έχουν τελικά και την ευθύνη να ε, καθιερώσουν τα FAB τα επόμενα δύο χρόνια και πρέπει να τους το θυμίσουμε αυτό. Όπως θα δείτε και στο έγγραφο που διένυμα, Σας έδωσα τα κριτήρια, τα πρώτα κριτήρια για τη δημιουργία των ΦΑΜ. Εγώ εξακολουθώ τώρα και επεξεργάζομαι ουσιώδη κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Πόσο δηλαδή καλά λειτουργεί το λειτουργικό τμήμα ενεργείου χώρου. Εγώ είμαι από τους παραδοσιακούς δικηγόρους. Γνωρίζω λοιπόν ότι μπορεί κανείς να κάνει μια θαυμάσια συνθήκη, αλλά χωρίς ουσία. Άρα ποια είναι η ουσία των ΦΑΜ, ώστε να σημειωθεί πραγματική πρόοδος και στη χωρητικότητα και στην ασφάλεια και στην ε, οικονομική αποδοτικότητα και στην φιλικότητα προς το περιβάλλον. Αυτή λοιπόν θα είναι η ατζέντα των ΦΑΜ και σε αυτήν θα προστίθεται και άλλα πράγματα, ουσιώδη κριτήρια και θα πούμε τότε το ΦΑΜ νούμερο 1 πληρεί το κριτήριο υπαριθμών 1, καλά τέλος πάντων ακόμη όχι, ώστε με την πάροδο του χρόνου να ε, δούμε πώς προχωρούν τα επιμέρους ΦΑΜ θα δείτε ότι έχουμε 9 FAB. Εγώ το σουηδικό και το δανέζικο τα θεωρώ ως πυρήνα ε, των μεγαλύτερων FAB. Αν είναι πράγματι έτσι λοιπόν θα έχουμε στο τέλος 8 μόνο συνολικά. Δύο εξ αυτών έχουν ήδη καθιερωθεί. Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και Σουηδικό και Δανέζικο. Έχουν λοιπόν καθιερωθεί επισήμω. Πρέπει να δούμε τώρα επί της ουσίας πώς λειτουργούν τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου. Ένα τρίτο FAB προχωρεί καλά. Αυτό λοιπόν που έχει και τον έλεγχο στην μεγαλύτερη κυκλοφορία είναι το της κεντρικής Ευρώπης. Στη σελίδα 8 θα κοιτάξετε. Είναι το κεντρικό λοιπόν αυτό FAB με την έννοια ότι έχει μέχρι και παραπάνω από 50% ε, της, ε, των κινήσεων. Μάλλον στις 2 Δεκεμβρίου θα υπογραφεί εδώ στις Βρυξέλλες η σχετική διακρατική συμφωνία και θα προβούν και σε δήλωση για το πώς προτίθεται να συνεχίσουν την συνεργασία αυτή γιατί αυτή η διακρατική συνθήκη λέει απλώς μόνον ποια, ποια όργανα θα είναι αρμόδια για να κάνουν τη δουλειά αυτά, αυτή. Θα πρέπει να δούμε μετά και το δεύτερο στάδιο ποιο είναι. Αυτό είναι το κεντρικό λοιπόν ε, λειτουργικό τμήμα ενεργείου χώρου. Ποια θα είναι τα ουσιώδη κριτήρια που πρέπει να επεξεργαστούμε. Θα σας αναφέρω λίγα για την ώρα. Το υπαριθμόν 1 είναι πώς διεξάγεται η συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, NSA στα αγγλικά, όχι National Security Agency, όπως ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά National Supervising Authority, εθνικές εποπτικές αρχές. Πώς συνεργάζονται λοιπόν στο FAB, Μπέκ που είναι Γαλλία, οι χώρες Μπενελούξ, Ελβετία και Γερμανία ε, και έχουν έξι εκπροσώπους. Αυτοί οι έξι αξιωματούχοι πώς συνεργάζονται. Υποτίθεται ότι θα έχει τη δυνατότητα ένα ΦΑΜ να έχει μία εθνική εποπτική αρχή. Ίσως να μπορέσει να γίνει αυτό. Πάντως η ιδέα είναι να είναι στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Δεύτερη ιδέα, στενή συνεργασία μεταξύ των παρόχων ε, εναέριας, ε, υπηρεσιών μάλλον εναέριας ε, πλοήγησης, αυτοί δηλαδή που κάνουν την πραγματική δουλειά. Πώς μπορούν να αναπτύξουν τη συνεργασία αποτελεσματικότερα. Τίθεται το θέμα λοιπόν της στενότερης συνεργασίας, όπως γνωρίζουμε από τις υπηρεσίες εναρίων μεταφορών συμμαχίες, η Γαλλία μάλιστα ε, θεωρεί ότι θα, θα, μπορεί να, έχει ένα, να υπάρχει ένας μόνο πάροχος υπηρεσιών για όλο το ΦΑΜΠΕΚ, το κεντρικό δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν συγχωνεύσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε το κάθε λειτουργικό τμήμα αερίου χώρου. Πώς εντατικοποιεί την συνεργασία, πώς γίνεται πιο αποδοτικό. Και όπως είπα πάντοτε για την ασφάλεια, την αυσυχωρητικότητα, ε, την αποδοτικότητα και την ε, φιλικότητα προς το περιβάλλον. Δεύτερο, η συνεργασία μεταξύ του στρατιωτικού, των στρατιωτικών αρχών και των πολιτικών αρχών. Σε ορισμένες χώρες όπως τη Γερμανία, οι πάροχοι εναερίων υπηρεσιών έχουν ήδη περιλάβει το στρατιωτικό τομέα. Επομένως, στου, στις αίθουσες ελέγχου ε, συνεργάζονται, είναι επιτόπου και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι συνεργάζονται με τους πολίτες. Αλλού έχουν ένα ε, πολιτικό ε, provider και ένα στρατιωτικό. Αλλά μην λησμονούμε ότι εμείς θέλουμε λιγότερη ρήπανση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στους εθέρες. Θέλουμε δηλαδή ένα αεροσκάφος το οποίο θα φύγει από το Α να πάει στο σημείο Β, να πάει σε ευθεία γραμμή και να μην αναγκάζεται να κάνει ζυξάκια να αποφύγει διάφορες ε, στρατιωτικές no-go areas. Μπορεί λοιπόν να, ε, να χωρίσουν και ε, χρονικά τις ε, υπερπτήσεις χώρων όπου δεν μπορούν να ύπτανται πολιτικά αεροσκάφη. Καμιά φορά το ζήτημα είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να λυθεί. Έχουμε και άλλα δύο κριτήρια που πρέπει να επεξεργαστούμε. Το πρώτο που λέγεται performance schemes. Η ιδέα αυτή ήταν αρχικά να δημιουργηθούν τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου, μετά όμως να ασκήσουμε πίεση στις χώρες και στις οργανώσεις να βελτιωθούν βάζοντας στόχους για την βελτίωση των επιχειρήσεών τους εξ αρχής, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε κατά πόσον η δημιουργία των FAB πραγματικά βοηθεί στη βελτίωση. Αυτά τα λοιπόν performance schemes μπορούν να γίνουν και σε εθνικό επίπεδο ή και ανά λειτουργικό τμήμα ενεργού χώρου που έχει περισσότερο νόημα εφόσον δηλαδή ιδρυθεί και οργανωθεί ένα FAB από κάθε άποψη να έχει και ένα performance scheme. Εργάζονται από αυτού οι χώρες μέλη, θα δούμε τώρα που θα καταλήξουν ώστε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος που επιθυμούμε να επιτύχουμε. Το τελευταίο ερώτημα είναι άλλωστε και μέσα στην νομοθεσία είναι και εκπληκτικό πόσα πράγματα περιλαμβάνει η νομοθεσία. Το τελευταίο κριτήριο είναι ότι η τελική ε, δημιουργία των ΦΑΜ θα πρέπει να αποδώσει μια προστιθέμενη αξία που να προκύπτει από την ανάλυση κόστου ωφέλους. Άρα δεν περνάμε τον καιρό μας διασκεδάζοντας, κάνοντας τη συνεργασία αυτή και την οργάνωση των ΦΑΜ. Όλοι το κοινό εν τέλει θα πρέπει να γνωρίζει για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά. Δηλαδή ποιο είναι το όφελος που προκύπτει υπέρ τη οικονομίας, υπέρ του επιβάτη, υπέρ του περιβάλλοντος. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι μονάχα η οργάνωση μιας διακρατική συνθήκης, αλλά να δούμε και πώ εκπληρούμε πραγματικά τους στόχους που φιλοδοξούμε να επιτύχουμε. Μέχρι τώρα και για λόγους χρόνου έχω συναντηθεί μόνο με τον Βέλγο και τον Γερμανό Υπουργό Μεταφορών. Η γυναίκα μου εξεράγει όταν είδε τι ε, εντολέ ε, αποστολών μου που περιλαμβάνουν δεν ξέρω πόσε πρωτεύουσε ε, χωρών Θύμωσε λοιπόν και μου είπε, μα τι κάνεις επιτέλους. Υποσχέθηκε λοιπόν, δεν θα πάω και στην τελευταία πρωτεύουσα, αλλά θα πρέπει να επισκεφθώ περισσότερες πάντως από αυτές που έχω επισκεφθεί ως τώρα. Έχω δει και τον Γενικό Διευθυντή της Eurocontrol. Η Eurocontrol είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην λησμονείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε, ε, συμβουλεύοντας την Eurocontrol, να χωρίσει τις θεσμικές διακυβερνητικές λειτουργίες από τις λειτουργίες προσφοράς υπηρεσιών. Και επειδή η ΕΑΣΑ, η European Air Safety Agency, ασχολείται κυρίως με τα θέματα της ασφάλειας και αυξάνει τις αρμοδιότητες της, ε, βασιζόμαστε στα δεδομένα που συλλέγει η Eurocontrol για λογαριασμό της Κομισιόν και δικό μας βέβαια του Κοινοβουλίου δηλαδή, και γι' αυτό συναντήθηκα με τον Γενικό Διευθυντή της Eurocontrol και με ε, την ε, ομάδα συνεργατών του που εργάζονται εξαιρετικά, που ε, είναι καλά οργανωμένοι, που μας βοηθούν πάρα πολύ. Πήγα να δω και την γερμανική υπηρεσία εναερίων ελέγχων. Θα ταξιδέψω λοιπόν και άλλο. Μην λησμονείτε πάντως ότι στόχος μου είναι να συνεργαστώ στενά και μαζί σας να ακούσω τις ιδέες σας, να μου εξηγήσετε τι θέλετε να επιτύχουμε, ποιοι είναι οι στόχοι δηλαδή που θεωρείτε ότι πρέπει να επιτύχουμε με τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου και τώρα με μεγάλη ευχαρίστηση να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Well, thank you, George, for that. George, ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα, για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. και βλέπω ότι ετοιμάζονται κάποιες ερωτήσεις. Ε, βεβαίως γνωρίζεις τις διαδικασίες σου, θα αρχίσουμε με τους, ε, τις διαδικασίες μας εδώ, ε, θα αρχίσουμε με τους συντονιστές. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Συντονιστά και σου εύχομαι καλή επιτυχία στην εργασία σου και πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και Βέβαια είναι το ενδιαφέρον ότι εμείς τώρα ρωτάμε και εσύ είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. και όπου η παρημιώδη ανυπομονησία σου να δούμε πώς θα σε βοηθήσει τώρα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε όντως στην θέση αυτή ένα πρόσωπο όπως ο Γιώργος Γιαρζεμπόσκι, διότι ήδη όταν βλέπουμε Δεκέμβριο 2012 ε, ανησυχούμε πραγματικά. Γνωρίζουμε πόσο αργά κινούνται τα γρανάζια των κρατικών μηχανισμών και ήδη ανησυχούμε. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και γνωρίζω ότι εσύ δεν ανέχεσαι τις καθυστερήσεις. Ε, γνωρίζουμε λοιπόν ότι και στις ε, εκθέσεις που θα μας υποβάλεις και πιστεύω ότι θα έχεις κατανόηση, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, να μας τα πεις καθαρά με το όνομά τους. Είμαστε μέλη μιας επιτροπής όπου συχνά ε, συζητούμε για διαθωτικά προβλήματα, προβλήματα υποδομών και δομών στις ε, χώρες μέλη και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αν κατάλαβα καλά από τα όσα είπες, για την ώρα έχουμε το πολύ δύο φαμπ τα οποία έχουν ξεκινήσει. Το τρίτο θα υπογραφεί τώρα τον Δεκέμβρη. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάποια κίνηση ή απολύτως καμία είναι ίσως υπερβολικά περίπλοκες οι προετοιμασίες. Δεύτερο, αυτό που είπες για την Eurocontrol, η κατανομή έργου, η κατανομή καθηκόντων μεταξύ ρυθμιστικού τομέα και παροχής υπηρεσιών είναι σημαντική και να παραμείνει. Θα πρέπει να τονιστεί. Μίλησες για στόχους και νομίζω ότι οι στόχοι αυτοί, δηλαδή αύξηση χωρητικότητα ή μάλλον βελτίωση τη ασφαλεια μείωση του κοστου κλπ, ε, προστασία του περιβαλλοντο οι στόχοι αυτοί μπορούν να είναι και αριθμητικοί. Όταν λέει κανεί, αύξηση της ωραία είναι. Αν πει κανεί όμως τριπλασιάζουμε τη χωρητικότητα, είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Συμφωνείς ότι μπορεί κανείς να περιγράψει ακριβέστερα τους στόχους, ώστε να έχει και τη δυνατότητα να ελέγχει καλύτερα του, την πλήρωση των στόχων από τη μια φάση στην άλλη. Επόμενο, αναφέρεται στον ρόλο ορισμένων διαρθρώσεων. Το ερώτημά μου εδώ είναι πώς βλέπεις το μέλλον και ποιο ρόλο θα παίξει η ΣΕΣΑ στο ε, χώρο αυτό. Και ποιες είναι, κατά τη γνώμη σου, οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που οφείλει να έχει η ΣΕΖΑ ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά της. Και μια τελευταία ερώτηση και μετά σταματώ. Το όλο αυτό σύστημα θα οδηγήσει και σε κάποια ανθρώπινα προβλήματα. Έλεγχη, δεν θέλω να ομιλήσω για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, αλλά το κόστος είναι ήδη υψηλό και θα γίνουν ακόμα, ακόμα υψηλότερο. Πού συζητείτε αυτό το θέμα ευθέως. Διότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους επαγγελματίες ώστε να εξευρεθούν οι καλύτερες λύσεις. Και νομίζω ο Belgo Control, ο οργανισμός δηλαδή εδώ, ο βελγικός, ε, θα είναι από τα πιο ακαθόδη θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλκαντράουι για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαζεμπόφσκι και να του πω ότι και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που τον ξαναβλέπω στις αίθουσε του Κοινοβουλίου και βεβαίως ευελπιστώ ότι στα επόμενα χρόνια θα τον βλέπουμε τακτικά και συχνά. Αυτή είναι μια πρώτη ε, συνάντηση, άρα ε, η, η, δεν χρειάζεται να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες, ε, αλλά μέχρι το 2012 θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Βεβαίως είμαστε όλοι θετικά διακείμενοι όσον αφορά την πρόταση αυτή και αυτό εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε, τόσο πιο καλά θα προχωρήσουμε. Όσο πιο αποτελεσματικά προχωρήσουμε, τόσο λιγότερα χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων θα δαπανίσουμε. Και όσο πιο γρήγορα ε, προχωρήσουμε, τόσο λιγότερες δαπάνες θα συνδέονται με τον έλεγχο της, ε, των, της εναέριας κυκλοφορίας. Μας ε, μιλήσατε για κάποια fabs τα οποία λειτουργούν ήδη και άλλα τα οποία προετοιμάζονται. Αλλά πέρα από τις ασκήσεις και τις προβλέψεις επί χάρτου, ε, το ζήτημα είναι τεχνικά, από τεχνικής απόψεως, πώς θα υλοποιηθούν τα φάμπς αυτά. Είπατε προηγουμένως ότι σε αυτά τα διάφορα FAB μπορεί η διαδικασία συντονισμού ή ολοκλήρωσης να διαφέρει από FAB σε FAB. Ε, ενδεχομένως λοιπόν να δημιουργηθεί ένα FAB το οποίο θα ε, υπερκαλύπτει το άλλο. Ε, η ερώτησή μου η συγκεκριμένη είναι θέλετε να επηρεάσετε, προτίθεστε να επηρεάσετε τη διαδικασία αυτή, θα ε, ε, εσείς θα προτείνετε κάποιο τρόπο ε, ε, έναντι κάποιου άλλου ή θα αφήσετε τα FABs να λειτουργήσουν μόνα τους και να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις γιατί είναι γεγονός ότι το κάθε ΦΑΜ θα προσπαθήσει να υλοποιήσει το δικό του σύστημα, αλλά δεν θα μπορούσε να ε, πάρει μαθήματα ε, και να ακολουθήσει παραδείγματα που λειτουργούν καλά σε διπλανά γειτονικά ΦΑΜ. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός, τέτοιου είδους συντονισμός ανάμεσα στα λειτουργικά τμήματα, έτσι ώστε να υπάρχει ε, πιο σίγουρη αποτελεσματικότητα, γιατί οι στόχοι είναι κοινοί ε, και επίσης για να ε, μπορούν να παρεμβαίνουν με κοινό και αποτελεσματικό τρόπο ε, σε κοινά προβλήματα όπως ας πούμε αυτό που αντιμετωπίσαμε με την ηφαιστειακή σκόνη. Ε, πώς θα γίνει λοιπόν μια αρμονική σχέση, η σχέση αυτή ανάμεσα στα FABs. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχήμα συντονισμού. Ποια είναι η άποψή σας. Έχουμε και τις τρίτες χώρες πέρα από τις FAB ε, που υφίστανται ήδη. Πώς ε, προτίθεστε να κινηθείτε. Τι επαφές θα έχετε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Έχετε μια ιδέα ήδη, έχετε κάποιο σχέδιο ήδη. Τελευταίο, μέσω της επιτροπολογίας υπάρχει ένα ε, ταμείο το οποίο μας επιτρέπει να εργαστούμε ε, σε ένα πολυετές πρόγραμμα. 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ε, και για τα ΦΑΜΠ προτίθεστε να συντονίσετε και αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο ε, θα εποπτεύεται τα ε, χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα μοιραστούν, θα κατανεμηθούν. Ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν σωστά και πιστεύετε ότι τα χρήματα αυτά αρκούν για τη δημιουργία των ΦΑΜΣ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Μαϊσνέρα από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας. Καλωσορίζω τον κύριο Γιαζεμπόφσκι. Ε, νομίζω ότι βεβαίως είσαστε πολύ άνετοι εδώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα των μεταφορών και αυτό είναι πολύ θετικό. Βεβαίως πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και το διαπιστώσαμε ε, με την περίπτωση του ηφαιστείου ε, στην ε, Ισλανδία. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού και επομένως χρειάζεται να δημιουργηθούν αυτοί, αυτά τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου, αυτά τα FABs. Πρώτη ερώτηση σε σχέση με το ηφαίστειο. Είχα τότε την αίσθηση ότι ότι η Ευρώπη δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη όσον αφορά την ασφάλεια να αντιμετωπίσει μια τέτοια ε, περίπτωση. Δηλαδή από το πιο απλό, ε, το να ξέρουμε εάν μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάξει ή όχι, ε, ε, ε, ήταν ερωτήσει στις οποίε δεν μπορούσε κανεί να απαντήσει. Επομένως, απαραίτητο ο συντονισμό όσον αφορά τα ΦΑΜ για αυτό το επίπεδο. Δεύτερον, υπάρχει στην Ευρώπη ο στρατιωτικός αναέριος χώρος και ο πολιτικός. Στην Γερμανία υπάρχει διασύνδεση. Απ' την άλλη μεριά χρήματα δεν υπάρχουν, τα ταμεία είναι άδεια και στη Γερμανία και στις άλλες χώρες. Επομένως δεν ήρθε η ώρα ε, να υπάρξει συντονισμός έτσι ώστε και τα χρήματα που δαπανώνται για να ε, διασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια των πτήσεων και των χώρων ε, δυνατότητας υπέρπτυσης να υπάρξει συντονισμός για αυτά. και υπάρχουν ε, πολλές πτήσεις οι οποίες ε, πρέπει να υποβάλουν αίτημα έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα, οι πέμπτες δεν αναφέρομαι απαραίτητα ε, σε μεταφορές επιβατών, αεροπλάνα δηλαδή που μεταφέρουν αλλά και μεταφορικά. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Επίσης, όσον αφορά τις άδειες, θα πρέπει συγκεκριμένα να ζητάμε άδειες. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Πιστεύω ότι εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. και βεβαίως ο ρόλος του θα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικός γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει στη δημιουργία των ε, ΦΑΜΣ, αυτών των λειτουργικών τμήματων εναερίου χώρου. Ερώτηση τώρα. Βεβαίως εγώ από κοντά παρακολουθώ τις εξελίξεις όσον αφορά τη δημιουργία ΦΑΠ στην Κεντρική Ευρώπη. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι ε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά είναι ε, συγκεκριμένοι. και με αυτούς θα πρέπει να συνεργαστείς και εσύ έτσι και αλλιώς. Είναι δύσκολο να αυτοσχεδιάσει κανείς ε, συνεργασία, αλλά πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι στο μέλλον η συνεργασία θα είναι πιο εύκολη. Πιστεύω ότι το θέμα της ε, στρατιωτικής, ε, της συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού αέριο χώρο είναι ε, πολύ σημαντικό θέμα. Γνωρίζουμε ότι μια καλύτερη, ένας καλύτερος συντονισμός, έστω και αν δεν φτάσουμε στη δημιουργία FAB, είναι ήδη ένα θετικό βήμα. και ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ήδη και στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί και έχουν συνεργαστεί σε μεγάλο βαθμό και επομένως ε, ε, ήδη, ήδη έχουν φτάσει σε κάποιους αρχικούς στόχους. Αλλά βεβαίως αν θέλουμε πλήρη κάλυψη τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Έγινε λόγος για μια νέα δομή. Ε, οι δικές μου καταβολές μου λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μόνιμο από το ε, πρόσκαιρο. Και επομένως δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε στις πρόσκαιρες λύσεις να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Ούτε θέλουμε όμως να αφήσουμε και τα πράγματα όπως έχουν τώρα και κάτι άλλο γενικής φύσεως. Βεβαίως οι εναέριες, οι, οι υπηρεσίες και οι εταιρείε που ασχολούνται με τις εναέριε μεταφορέ θέλουν να αυξήσουν όσο γίνεται περισσότερο ε, την εργασία τους. Εάν όμως υποθέσουμε ότι το FAB έχει σαν στόχο και την εξοικονόμηση, την μείωση των ε, εκπομπών και των ε, ρήπων, ε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουμε νέου, νέες έχουμε νέους κινητήρες, έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις, το πρόβλημα παραμένει και διαρκώς θα αυξάνεται και βεβαίως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μειωθούν οι εκπομπές όταν λέμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε την εναέρια κυκλοφορία, όταν, θέλουμε να, όταν ήδη από τώρα λέμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε ε, τις εναέριες ε, μεταφορές. Uh, Ευχαριστώ. Σε αυτό τον πρώτο γύρο των συντονιστών θα δώσω το λόγο στην κυρία Τσάκη Φώστερ για τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώ ήρθε, Τζόρτζ. Εγώ ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφευγε ήρεμα και θα συνταξιδοτούσαν. Δεν με εξέπληξε καθόλου λοιπόν η ανάμειξή σου στα λειτουργικά του μεταναέριου χώρου. Εμείς ήμασταν υπέρ του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και οι περισσότεροι από εμά είμαστε άνθρωποι πολλά χρόνια στην πολιτική και φεύγουμε, ξαναρχόμαστε και βλέπουμε με ικανοποίηση πόσο έχουμε προχωρήσει και πόσο έχουμε προοδεύσει. Γιατί όλα αυτά που είπες για τη συμφόρηση, για τη χρήση του εναέριου χώρου που έχουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με πιο φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, με πιο αποδοτικό τρόπο και για την βιομηχανία. Όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερες ε, ήταν θέματα που για πολλά χρόνια υποστήριζαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ εκφίσως είμαι αισιόδοξη και μάλιστα οφείλει κανεί αν είναι ευρωβουλευτή, να είναι και αισιόδοξο. Αλλά Είπε έχουμε εννέα τέτοια φαμπ, έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, ήδη ένα-δυο φαμπ λειτουργούν. Μπορεί να έχουμε ένα MOU και να συμφωνήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα κολλησιεργήσουμε. και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για σένα. Είχαμε το πρόβλημα της ηφαιστειακής ε, τέφρας ε, το καλοκαίρι και τότε όλοι καταλάβαμε πόσο επίγον είναι το θέμα και ότι θα πρέπει να συντονιστούμε, αλλά υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να διαθετηθούν. Και είναι και θέμα των κρατών μελών. Και δεν ξέρω πώς ε, η Κομισιόν μπορεί να, να πιέσει τα κράτη-μέλη για να προοδεύσουν. Έχουμε και δύο άλλους τομείς. Έχουμε τα διάφορα συμφέροντα δεν είναι ότι θέλουμε να απολυθούν ε, ε, ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές στις αμοιβέ μεταξύ των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας και φυσικά θέλουν να κρατήσουν τις θέσεις τους οι άνθρωποι, αλλά μιλούμε για ένα είδος ε, ενοποίησης της χρήσης του ενέργειου χώρου. Και αυτό είναι και ο γενεσιουργός λόγος των FABs. Η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στη χρήση του ενέργειου χώρου. Επίσης, η συνεργασία πολιτικής στρατιωτικής αεροπορίας. Ιστορικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε ελαστική χρήση του ενέργειου χώρου. Δεν είχαμε πρόβλημα ε, με τα ΦΑΜΠ, όπως συνέβη στην Γερμανία, για παράδειγμα. Τι γίνεται όμως με τα άλλα κράτη-μέλη ό,τι αφορά το διαχωρισμό ή χρήση του αερίου χώρου από την πολιτική και τη στρατιωτική αεροπορία. Βέβαια, δεν μπορούμε να δούμε ξεχωριστά τα ΦΑΜ. Είναι θέμα και ΣΕΖΑ. Υπάρχουν τεράστιες δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Ήδη έχει προβλεφθεί κάποιος προϋπολογισμός. Αλλά αυτοί που θα υποβάλουν τις τεχνικές λύσεις μέχρι στιγμής καθυστερούν κάπως. Αλλά έχουμε και τις επενδύσεις από τη ΣΕΖΑ που είναι προσχέδιο προπολογισμού, στο προσχέδιο ακόμη προπολογισμού, θέλουν κάποια ενημέρωση και για τα οικονομικά. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι με τις ερωτήσεις τους, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου, κολοσιαίο έργο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αναποφασιστικότητα έλλειψη βούληση, αλλά είναι και θέμα κρατών μελών. Και παρά τα δημοσιονομικά ζητήματα που είναι διακρατικά, θα πρέπει να γίνουν και σημαντικές αλλαγές. Τώρα, ε, τι μπορείς να κάνεις εσύ ως συντονιστής και πώς μπορείς να προωθήσεις το θέμα αυτό και με τους συνομιλητές σου και στις συναντήσεις που θα έχεις. Έγιναν πολλές καθυστερήσεις το 2010. Δεν μπορούμε να έχουμε επανάληψη της ηφαιστειακής τέφρας. Εγώ έχω, είχα 25 χρόνια πείρα στον κλάδο αυτό και πρώτη φορά είδα τέτοια κακή αντιμετώπιση ε, τόσα αεροπλάνα εγκλωβισμένα και καθυλωμένα σε αεροδρόμια και τόση κολυσιεργία. Τέτοια καταστροφή δεν είχαμε δει, είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να βελτιωθεί η κατάσταση και με τη Eurocontrol και με τα, τη σύσταση των FAB. Περιμένω λοιπόν το σχολιασμό σου και τις απαντήσεις σου σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Τζάκη. Γιώργ, θέλει να απαντήσει ερωτήσει στο συντονισμό και να αφήσουμε του υπόλοιπου έξι ομιλητέ για το δεύτερο γύρο των ερωταπαντήσεων. Περιμένουμε τι απαντήσει από τον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις διάφορες ερωτήσεις και να δώσω κοινέ απαντήσεις. Όντως είμαι ανυπόμονος άνθρωπος αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαι και διπλωμάτης, ε, να δείξω μια διπλωματικότητα, να συζητήσω με όλους. Δεν μπορώ να σπέβδω και να εκφέρω την προσωπική μου γνώμη για την κατάσταση. Δεν θα ήταν ε, fair, δεν θα ήταν δίκαιο κάτι τέτοιο, ούτε θεμητό. Δεν μπορώ να παρουσιάζω τις δικές μου ε, απόψεις. Χρημάτισα και δικαστή ένα διάστημα και ξέρω ότι πρώτα πρέπει να ακούει κανεί του άλλου και μετά να διαμορφώνει γνώμη. Συναντήθηκα με πολλούς ε, διευθυντές ε, και το έργο τους είναι εξαιρετικό, αλλά αυτή τη στιγμή όλα σχεδόν εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και μόνο με έναν τρόπο μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, με συνομιλίες, με συναντήσεις με πολλούς, ε, να δώσουμε κίνητρα στα κρατημέλη, να τα παροτρύνουμε και να ασκήσουμε και μία ελαφριά πίεση. Και φυσικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιέσει όσο μπορεί. Και αν δεν τηρηθεί η προθεσμία του 2012, φυσικά έχουμε και τα 11 μέσα κατά των ε, κρατών μελών για παραβίαση των προθεσμιών της συνθήκης. Οπότε προς το παρόν θα δώσουμε κάποια κίνητρα, κάποια ενάσματα, θα προσπαθήσουμε να θαρρύνουμε και να τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και θα δούμε. Αυτή τη στιγμή η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είναι καλό και τι λιγότερο καλό. Και όσοι έχουν επαφές με τις κυβερνήσεις θα πρέπει να τις αξιοποιήσουν για να προωθήσουν αυτό το θέμα. Προσπαθήστε να δείτε στις χώρες σας πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση είναι καλή. Τώρα, για τα τεχνικά ζητήματα δεν πρέπει να είμαστε ε, υπερβολικά βιαστικοί. Το ΣΕΖΑ είναι πολύ σημαντικό. Σε δύο εβδομάδες θα έχω συνεδρία, συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΣΕΖΑ και φυσικά ε, χρειαζόμαστε το ΣΕΖΑΡ αλλά χρειαζόμαστε και τα FAB. Και όταν θα έχουμε, θα περιμένουμε τα πρώτα προγράμματα και τον εξοπλισμό του ΣΕΖΑΡ. Και μην ξεχνάτε και το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, δίνει κονδύλια στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Βέβαια δεν μπορώ να τα πω όλα έξω από τα δόντια στα κράτη-μέλη, οπότε τι μπορώ να, να πω. Χρειαζόμαστε το ΣΕΖΑΡ για την πραγματοποίηση των ΦΑΜ. Όχι, τα ΦΑΜ μπορούμε να τα ε, πραγματοποιήσουμε και χωρίς το ΣΕΖΑΡ. Γιατί να περιμένουμε το ΣΕΖΑΡ μπορεί να περιμένουμε 10 και 20 χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρουν συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα μπορέσουμε να καταμετρήσουμε την πρόοδο και την εξέλιξη. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τέτοια κριτήρια και έχουμε μονάδες ε, και σώματα που προσπαθούν να καταμετρήσουν αυτή την πρόοδο. Καταρτίζονται και εκθέσεις, λαμβάνουμε γνωμοδοτήσεις, αλλά αντίστοιχη ευθύνη έχουν και τα κράτη-μέλη. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καταλήξουν σε κάποια θεμελιώδη κριτήρια. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Συντονιστής δεν μπορούν να υποχρεώσουν τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επεξεργαστούν τα ποσοτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και να ενημερωθούμε για τα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά τα ισχύοντα FAB θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο όντως είναι λειτουργικά, κατά πόσο προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία και αν όντως υπάρχει προστιθέμενη αξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα FAB ως παραδείγματα προς μίμηση. Δεν θα πρέπει να έχουμε φαμπ με διαφορετικές αποδόσεις, ορισμένα να είναι πιο αποτελεσματικά και άλλα λιγότερα. Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να καθορίσουμε κάποια κριτήρια για την καταμέτρηση της πρόοδου και να περάσουμε κατόπιν στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας των φαμπ. Τα κράτη-μέλη θα είναι ανέκαθεν αρμόδια για τα θέματα αυτά. Βέβαια υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα και κάθε χώρα ε, υιοθετεί την οργάνωση που κρίνει σκόπιμη. και σε άλλες ε, χώρες έχουμε εποπτικές αρχές, σε άλλες χώρες ε, το ίδιο το Υπουργείο αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα. Επίσης έχουμε δεύτερο επίπεδο που είναι τα εθνικά σώματα ελέγχου και το τρίτο επίπεδο που είναι ο πάροχος υπηρεσιών αρμόδιος για την εναέρια ασφάλεια. Και φυσικά χρειαζόμαστε κάποιες κοινέ πρωτοβουλίες και κάποια κοινά προγράμματα. Και αν έχουμε FAB, στα οποία συμμετέχουν περισσότερες χώρες, τρεις, τέσσερις, πέντε, κάθε χώρα θα έχει φυσικά τη δική της έδρα που θα αναλαμβάνει την ενέργεια ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και συνεργασία ό,τι αφορά την κοινή κατάρτιση των ελεγκτών. Θα πρέπει να πάει στην να λαμβάνουμε υπόψη σε διάφορα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Στην Γαλλία έγιναν αρκετέ απεργίε. Δεν να τις κατακρίνω φυσικά. Ούτε θα πρέπει να μειωθούν οι θέσεις απασχόλησης ή να δεχθούμε ένα dumping στις αμοιβέ των ελεγκτών. Θα πρέπει όμως να αξιοποιήσουμε καλύτερα ε, τα προσόντα και να προσλάβουμε ελεκτές ενέργειες κυκλοφορίες, γιατί μας λείπουν ε, υπάλληλοι. Και μάλιστα και στο σιδηροδρομικό πακέτο είχαμε αντίστοιχα προβλήματα με λοιπές προσωπικό. Θα προσπαθήσω πάντως με κοινωνικό διάλογο να θέσω τα θέματα αυτά, ώστε να μην προκύψουν αντίθετες κινήσεις, αντιστάσεις που ίσως είναι αδικαιολόγητες. Δηλαδή μόνο χωρίς να έχει δηλαδή υπάρξει πρώτα Τώρα για την interconnectivity δεν είναι δυνατόν το ένα FAB να βάζει τους αεροδιαδρόμους σε αυτό το ύψος και το επόμενο να τους κατεβάζει σε αυτό το ύψος. Ε, είναι δύσκολο το θέμα. Πρέπει να συζητήσουμε τίσουν και τα ΦΑΜ μεταξύ τους και με τους στρατιωτικούς που για παράδειγμα υπάρχουν ε, κάποια ε, τμήματα της επικράτειας όπου δεν μπορεί να ε, γίνει πτήση πολιτικού αεροσκάφους διότι είναι no-go areas, είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Γνωρίζετε ότι αυτό το, με αυτό επιφορτήσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάξει μέχρι τέλους του έτους ένα δίκτυο του management. Είπαμε ότι το Eurocontrol ή κάποια άλλη αρμόδια οργάνωση, μάλλον αυτή όμως θα είναι, λόγω και της εμπειρίας δεκαετιών, έχουν και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, έχουν και τη μεθοδολογία εργασίας. Περί αυτού πρόκειται, δηλαδή πώς θα οργανωθεί καλύτερα ο αέριος χώρος και πέραν των FAB και στην βάση αυτού του δικτύου management. Ελπίζω ότι θα έχει κρυθεί το θέμα μέχρι τέλος του έτους και θα μπορέσει να αρχίσει συνεργασία. Σε ό,τι αφορά συνεργασία στρατιωτικού και πολιτικού τομέα και, τα, και τους σχετικούς φορείς. Είναι διαφορετική κατάσταση από χώρα σε χώρα. Και καμιά φορά με πολύ παθιασμένη στάση και των στρατιωτικών και των ε, πολιτικών φορέων. Θα δω τώρα με τον διάλογο πώς θα προχωρήσει. Χρειάζεται προσοχή ε, να μην, όπως είπα, προκύψει κάποια αντίσταση. Οι χώρες μέλη βεβαίως έχουν την κυριαρχία. Γνωρίζω ότι η Ισπανία, για παράδειγμα, είναι πολύ, ε, πώς να πω, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να διατηρήσει απολύτως την κυριαρχία. Δεν θέλουμε να εξοργήσουμε τους Ισπανούς, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Αλλά σε τελική ανάλυση πρέπει να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε. Εσεί, κυρία Λίχτενμπέργκερ έχετε δίκιο που λέτε ότι εάν υπάρχουν, υπάρχει περισσότερη κυκλοφορία θα υπάρχουν και περισσότερες εκπομπές ρήπων. Ο καθήκον μας δεν είναι να ανακόψουμε την πορεία των αερίων μεταφορών, αλλά να την οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι εάν όντω οργανωθεί καλύτερα, θα έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα και από άποψη ρήπων. Δεν ξέρω αν θα επιτύχουμε 12% μείωση εξαρτάται από το ποιον προσανατολισμό θα λάβουμε. Βλέπω ότι μακρηγόρησα αρκετά. Ίσως έχω λησμονήσει κάτι σημαντικό. Αλλά πάντως ρωτήστε με ή αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο αργότερα ή στείλτε μου ένα email. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα για το 2012, μέχρι το 2012, και στο Συμβούλιο των Υπουργών αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά νομίζω θα γίνεται μια ενδιάμεση έκθεση και θα την συζητούμε. θα σας ε, πω για δύο τομείς που με απασχολούν ιδιαίτερα. Το κεντρικό ευρωπαϊκό ΦΑΜ και όλος ο σχετικός προβληματισμός με την πρώην Ιουκοσλαβία, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο, δύσκολο όπως είπατε και εσείς. Ωστόσο είναι σημαντική η αεροδιάδρομη αυτή, προσφέρουν και τη διασύνδεση με την Ελλάδα και την Κύπρο, άρα πρέπει να γίνει. Το, το Med, αυτός ο τομέα είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολος. Το συντομότερο δυνατόν θα έλθω σε επαφή με τον Ιταλό Υπουργό Μεταφορών. Πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, οι εμπειρογνώμονε, έχουμε πραγματικά σε όλα τα επίπεδα εξαιρετικού εμπειρογνώμονε και στην Κομισιόν και στην Ευρωκοντρόλ και στι εθνικέ αρχέ. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Θέλουν οι χώρε μέλη πραγματικά να εγκαταλείψουν κάποιες απειρχιωμένες μεθόδους, θέλουν όντως να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, θέλουν να συζητήσουν για νέες μεθόδους. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συζήτηση με τις χώρες μέλη, κομισιόν και χώρες μέλη. Ας συνεργαστούμε λοιπόν έτσι περαιτέρω και βλέπουμε. Ευχαριστώ για τον πρώτο αυτό γύρο. Έχω 7 εγγεγραμμένους για τον δεύτερο γύρο, ο κύριος Πάσπα. Πασπά. Bienvenido, Jorge, a Καλώς ήρθες, Χόρχε, στην Επιτροπή σου. Εγώ ξέρω ότι... Ε, επειδή είσαι καλός άνθρωπος, παρόλο που έχεις κακό χαρακτήρα, σίγουρα θα πας στον παράδεισο. Αυτό είναι ε, παρηγοριά για τους αγνωστικιστές. Γιατί οι χριστιανοί ξέρουν ότι πάνε κατευθείαν στον παράδεισο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες που αναφέραμε, που ακούσαμε, η φυσική τέφρα και η κρίση που ακολούθησε ήταν απόδειξη της ανικανότητας της Ευρώπης, αλλά όχι μόνο. Γιατί η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός, δεν θέλουμε να επιρρύψουμε ευθύνε. Απλώς διαπιστώνουμε τις αδυναμίες. Στην Ισπανική Προεδρία καταλήξαμε σημαντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και φυσικά θα πρέπει να εγκομιάσουμε ε, το έργο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνέβαλε τα μάλα στη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Ε, τι γνώμη έχεις εσύ για τη συμφωνία αυτή, πώς την αξιολογείς και επίσης ε, ένα σημαντικό τμήμα ε, του Ατλαντικού και ε, τη Λατινική Αμερική θα την αφήσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετέχουμε και εμείς στη λήψη των αποφάσεων και σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ κυρία Τσικάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας ευχαρώ, κύριε Γεζομπόφσκι για την ε, νέα θέση και τα νέα σας καθήκοντα. Τον Ιούλιο δημοσιεύθηκε ένας κανονισμός ό,τι αφορά τα κριτήρια επιδόσεων για τα FAB. Αργότερα λήθησαν κάποιες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και δόθηκαν κονδύλια για την σύσταση ορισμένων φαπ Πώς θα υλοποιηθεί όμως ο συντονισμός, γιατί χρηματοδοτήθηκαν και κάποια προγράμματα που δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια επιδόσεων, γιατί τότε δεν υπήρχαν κριτήρια επιδόσεων. Οπότε ρωτώ πώς ε, θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα ΦΑΠ. Μια και ο κανονισμός ε, δημοσιεύθηκε μόλις τον Ιούλιο. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο συντονισμού για την ίδρυση των ΦΑΠ. αλλά και τη μελλοντική χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020. Ελπίζω να υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγηση και βελτίωση για τι επόμενε χρονιέ. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβλέπω τον κύριο Γεζαμπόφσκι και θυμάμαι την καταπληκτική μας συνεργασία στις αρχές της δεκαετίας του 90 και τις πολυάριθμες συναντήσεις που είχαμε με το Συμβούλιο και τον Γκίντερ Λουκ που διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο τότε στις διαπραγματεύσεις. Επανερχόμαστε στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να έχουμε μια γενικότερη επισκόπηση να δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία και με απόσταση και να δούμε τα περίπλοκα σημεία και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί υπάρχουν πολλά καθόδη ζητήματα και δυσεπίλητα. Τα γνωρίζουμε, αλλά εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε θα έχουμε επαφέ με τις εθνικέ κυβερνήσει και τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να σας διευκολύνουμε, να σας βοηθήσουμε να βγούμε από το διέξοδο. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα κρεμή προβλήματα, ποια είναι τα πιο δυσεπίλητα θέματα και να μας πείτε πότε θα δώσετε το πράσινο φως ή μερικές φορές αν ανάβει πορτοκαλί ή κόκκινο. Σε ό,τι αφορά το Net Fab της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πώς θα λειτουργήσει. Χώρες όπως ε, η Αλβανία, η Αίγυπτος, ε, ακόμη και η Ορδανία που έχει καθεστώς παρατηρητή, πώς θα συνεργαστούν και ποια είναι η θέση του Ισραήλ στο λειτουργικό τμήμα αέριου χώρου της ε, νότιο-ανατολικής Ευρώπης και Και η θέση του Ισραήλ στο ΦΑΜ αυτό, ποια θα είναι. Κύριε Γεσεμπόλς, και φυσικά δεν θέλω να επέμβω στην ε, ιδιωτική σας ε, σφαίρα, στην προσωπική σας ζωή, αλλά πραγματικά κατανοώ την ε, γυναίκα σας και τα, το θυμό της, αλλά εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας και μπορείτε να υπολογίσετε σε εμάς και για την ασφάλεια του γάμου σας, αλλά και για την ασφάλεια του ενέργου χώρου, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η ζωή που θα έχετε ως συντονιστής θα σας δημιουργήσει προβλήματα στη συζυγική σας ζωή. Α, δεν ήξερα κύριε Βαντάλεν ότι είστε και σύμβουλος γάμου. Ο κύριος Φιντάντσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, εγώ δεν έχω τις θαυματουργές ε, ιδιότητες ε, του κύριου Βαντάλεν. Θα ήθελα απλώς να ευαθύνω στο θέμα του Blue Med. Γιατί στους πίνακες και τα έγγραφα που μα ο συντονιστής υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Το μόνο FAB που έχει κενά σημεία είναι το FAB Blue Med. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εκεί, είναι κενά όλα τα τετραγωνίδια και πέραν των όγκων κυκλοφορίας, του όγκου κυκλοφορίας που μας υποχρεώνει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο FAB, γιατί έχουμε πάνω από 50% της ενέργειας κυκλοφορίας στο FAB της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το FAB Blue Med, που έχει και ιδιαιτερότητα αλλά και στρατηγική σημασία, γιατί είναι το μόνο ΦΑΜΠ που καλύπτει ένα αέριο χώρο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει στρατηγική σημασία και για τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρώπης, γιατί ενδιαφέρει τη Μεσόγειο, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, εκτός από την Ευρώπη. Υπάρχουν ακόμα όμως ε, τεράστιες δυσκολίες ό,τι αφορά την ε, ε, υλοποίηση των φιλοδοξιών μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και δεν ξέρω κύριε συντονιστά πώς μπορείτε να παρέμβετε εσείς για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς σε αυτό το FAB. Και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα αναθεωρήσουμε τις προθεσμίες που από ό,τι φαίνεται είναι αδύνατον να τις ατηρήσουμε. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπουμε στην Επιτροπή μας, κυρία Γιαζεμπόφσκη. Και ευελπιστώ ότι θα φέρετε σε αίσιο πέρας τα καθήκοντά σας ως συντονιστού των ΦΑΜ και θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον πολυπόθετο στόχο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Η επίκριση που ασκείται κατά τον ΦΑΜΠ και από πολλά κράτη-μέλη είναι ότι είναι άχρηστα. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεπεράσουν ένα ψυχολογικό φραγμό προκειμένου να συνηθίσουν στην ιδέα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Και είναι πολύ καλό που αρχίσαμε τις συζητήσεις για τα FAB, αυτά τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου. Θα εξετάσουμε κάποια κριτήρια επιδόσεων, γιατί ήδη υπάρχει δίκτυο οδών, το οποίο έχει αναλάβει Eurocontrol, αλλά αυτό που θα πρέπει να, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για τα FAB είναι ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας. Κυρίως αποτελεσματικότερο έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας. Και αν έχουμε κέντρα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε στις πιο αποτελεσματικές θέσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ελέγχους, σημεία ελέγχου και στις δύο πλευρές των συνόρων, σε γειτονικέ περιοχές. Στο μέλλον μπορούμε να το καταργήσουμε από τη στιγμή που θα έχουμε FAB. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένθεν και ένθεν κέντρα ελέγχου στα FAB. Υπάρχει ένα άρθρο του κανονισμού που λέει ότι τα FAB θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους κατά την το προσδιορισμό σημείων ελέγχου. Αναρωτιέμαι λοιπόν πως θα πρέπει να υποβληθεί μία πρόταση για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Μία πρόταση για σημεία ελέγχου στην Ευρώπη με βάση τον, Ευρωπαίο, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Η φιλοσοφία δηλαδή αυτή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Νομίζω ότι αυτό είναι το, και το πιο σημαντικό που θα πρέπει να κάνουμε στα FAB. Και άλλα θέματα είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα για να γίνουν όντως λειτουργικά τα FAB και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται σε αυτό που είπε η συνάδελφος για το ΣΕΖΑΡ. Το ΣΕΖΑΡ για την φάση ανάπτυξης σημείο φετηρίας τον Ιανουάριο του 2014. Είναι προφανές λοιπόν ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, το ελπίζω, η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να στηρίζεται στη διάρθρωση του, του, της ενέργειας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και όχι στα ΦΑΜΠ. στη διάρθρωση ελέγχου των ΦΑΜΠ. Και αυτός ο χάρτης με τα σημεία ελέγχου είναι πολύ σημαντικό και αυτό απασχολεί τους όσους ασχολούνται με το ΣΕΖΑΡ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνεργασία ΣΕΖΑΡ και ΦΑΜ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, μακάρι να τηρήσουμε την προθεσμία του Δεκεμβρίου 2012, κατά τη γνώμη μου είναι λίγο τοπικό. Σας ευχαριστώ κύριο Σκούν. Εδώ είμαι Γιώργ. Χαίρομαι που ένα πρόσωπο με τη δική σου γνώση, τη δική σου ανυπομονησία και το δικό σου γοητευτικό χαμόγελο, αναλαμβάνεις καθήκοντα συντονιστού και θα θα συμπαραστέκεσαι, ας το πω καλύτερα, ε, στην προσπάθεια του Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ θεωρώ επίσης σημαντικό να συνεργαστεί κανείς στενά και με τις χώρες μέλη. Εκεί θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο το που μπορούμε να επιτύχουμε κάποια οικονομικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα οι κοινέ προδιαγραφές. Δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι θα εργάζονται στον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας να έχουν την ίδια εκπαίδευση. Επίσης, το λογισμικό. Εκεί μπορεί να γίνει σημαντική εξοικονόμηση, εξοικονόμηση κλίμακος και βεβαίως να υπάρχει και συμβατότητα για την ασφάλεια στους εθέρες. Όχι μόνο να έχουμε ένα ενίο απελευθερωμένο οικονομικά ενέργειο χώρο. Είμαστε ταυτόχρονα υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβατών. Επίσης η συνεργασία με τους στρατιωτικούς. Βαντάλεν είπε τι γίνεται με την Ιορδανία και το Ισραήλ θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις αρκετά το γοητευτικό σου χαμόγελο και απέναντι στους πιλότους των ε, τουρκικών μαχητικών που μπαίνουν στον ελληνικό ενέργειο χώρο. Και μια ερώτηση. Πρόσφατα συζητήσαμε την έκθεση της κυρίας Ντεβεράκ για ατυχήματα και συμβάντα στον ενέργειο χώρο. Και εκεί παίζουν σημαντικό οι εθνικές αρχές, σημαντικό ρόλο οι εθνικές αρχές και σε ό,τι αφορά την συνεργασία και σε ό,τι αφορά την διασύνδεση των εθνικών αρμοδιοτήτων. Πάλι παίζουν όμως εδώ ρόλο στην ασφάλεια. Και για την ασφάλεια των εθέρων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πώ θα φροντίσει ώστε να υπάρξει συνεργασία και σε αυτά τα δεδομένα. Σε σάδα. Ευχαριστώ. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι πραγματικά ανεκτήμητη πρωτοβουλία και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι ε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει υψηλό κόστος, ε, αύξηση των αεροπορικών μεταφορών και όλοι είμαστε υπέρ, αλλά δεν ξέρω αν ε, η δημιουργία των 9 FAB είναι ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός ή όχι ακόμη. Έχω λοιπόν μία σύντομη και απλή ερώτηση. Πότε θα είναι το επόμενο βήμα, γιατί αυτά τα εννέα φάμπ είναι μεταβατική φάση. Κάποια στιγμή θα έχουμε τον, Ευρωπαίο, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Σε ποια φάση βρισκόμαστε όμως. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν χαμηλότερο κόστος, αλλά και λιγότερους ελέγχους ενέργειας κυκλοφορίας. Εμείς έχουμε περισσότερους ε, ελέγχους. Τι γίνεται με τους ε, ελέγχους, γιατί ε, θα έχουμε και τη συνάντηση με τους ελεγκτές των Βρυξελών. Γιατί είναι σημαντικό θέμα το προσωπικό των ελεκτών ενέργειας κυκλοφορίας. Και μία άλλη ερώτηση γιατί έχετε συναντηθεί με πολλούς πολιτικούς. Ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτού του, του σχεδίου, ποια είναι τα προσκόμματα, γιατί λέμε ότι μέχρι το 2012 ούτε το πρώτο βήμα δεν θα έχουμε ολοκληρώσει. Ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι η κίνδυνη, ποια είναι τα προσκόμματα, τι εμποδίζει στο μέλλον να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάβεσα. Δεν έχω εστονική μετάφραση σήμερα και γι' αυτό θα προσπαθήσω να πω τις σκέψεις μου στα αγγλικά. Και εγώ λοιπόν ε, ε εκφράζω το καλωσόρισμα στον ε, κ. Ζεμπόσκη. Τώρα η ερώτησή μου. Είπε ότι δεν μπορεί να επιτύχει τόσο γρήγορα. Ποια είναι τα προβλήματα ή ερωτήματα γιατί δηλαδή δεν επιτυγχάνουν οι χώρες μέλη τόσο γρήγορα να προχωρήσουν σε αυτό το θέμα. Είπατε ότι θα επισκεφτείτε τις χώρες μέλη. Τι είδους απαντήσεις αναμένετε να λάβετε από ε, τις χώρες μέλη. Είναι περισσότερο η έλλειψη πόρων, είναι περισσότερο η έλλειψη της πολιτικής ε, βουλήσεως, είναι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ εταιριών, αεροδρομίων και ούτω καθεξής. Ο κύριος Βαντάλεν έδωσε μια καλή συμβουλή. Πώς ε, δηλαδή, τι κίνητρα να προσφέρετε στη σύζυγό σας και εν τέλει τι έχετε ε, στη διάθεσή σας ώστε να παρακινήσετε και τις χώρες μέλη. Έχετε κάποιες ιδέες. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη, λέει η κυρία Μάισνερ, πράγματι. Ένα συνάδελφο τη ομάδα μου που αναγκάστηκε να φύγει από την αίθουσα μου έδωσε μια ερώτηση. Ένας από τους στόχους της βελτίωσης δηλαδή του περιβαλλοντικού αντικτύπου είναι και αυτό ένα θέμα μεγάλο. Τι μπορεί να γίνει για την μείωση των ρήπων. Ταυτόχρονα έχεις βάλει ω στόχο και την αύξηση τη χωρητικότητα των εθερών. Άρα δηλαδή μήπως η μία προσπάθεια ακυρώνει την άλλη. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει πιο συγκεκριμένα ο συντονιστής των ΦΑΜ ώστε να επιτύχει μεγαλύτερη, ε, πιο φιλικό χαρακτήρα προς το περιβάλλον. Πολύ σύντομα θα παρακαλέσω να απαντήσεις, αλλά πρώτα θα ήθελα να κάνω και εγώ ορισμένα σχόλια. Νομίζω ότι ε, δημιουργήθηκε η αίσθηση και από τα λεγόμενα των συναδέλφων ότι μας απασχολεί το θέμα του Σεζάρ. Βεβαίως μπορεί κανείς ε, να ανταπαντήσει ότι ε, ότι εάν το ηφαίστειο της Ισλανδίας δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην ευρωπαϊκή ε, αεροπορία ενδεχομένως να ε, είναι και κάτι καλό, ε, διότι στην ουσία πυροδότησε μια πιο έντονη συζήτηση ε, γύρω από τα θέματα της πολιτικής αεροπορίας και οι ίδιες οι εταιρείε, αλλά και οι απλοί πολίτες άρχισαν να αναρωτιούνται και να ρωτούν τι θα γίνει, προχωράμε καθόλου για την ενοποίηση του εναέριου χώρου, προχωράμε καθόλου όσον αφορά τα ΦΑΜΠ και τα ΦΑΜΠ επομένως είναι μια απάντηση σε αυτή αυτήν την ε, ε, ανησυχία ε, κατά κάποιο τρόπο πίεσε τα κράτη να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν θα επιλέξουμε το Σεζάρι ή τα ΦΑΜΣ ή τα ΦΑΜΣ και όχι τα Σεζάρι, οτιδήποτε. Το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε. Και η άποψη του κυρίου Ασάντο είναι ενδιαφέρουσα βλέπουμε ε, την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, βεβαίως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς ίδια. Από τη μία πλευρά έχουμε 21 αρχές για 18 εκατομμύρια πτήσεις και από την πλευρά της Ευρώπης έχουμε 47 ε, παρόχους ε, αεροπορικών ε, μεταφορών και νομίζω ότι και από αυτό μόνο καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα και το μέγεθος του προβλήματος το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Θα θυμάσαι φαντάζομαι George ότι όταν πουλήσαμε εντό εισαγωγικών την ιδέα αυτή με την Κομισιόν το, πριν από πάρα πολλά χρόνια και είχε έρθει εδώ και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ο οποίος ε, μας πούλησε ας πούμε την ε, ιδέα αυτή και μας είπε ότι ε, ήταν εξαιρετική ιδέα και ότι θα γίνει αποτελεσματικότερη η ενέργεια κυκλοφορία και ένα από, τη, τα πλεονεκτήματα θα ήταν ότι δεν θα περιμένανε, δεν θα υπήρχαν αυτά τα σλότ στα αεροδρόμια και αεροδρόμια τα οποία να περιμένουν ε, ώρες πριν απογειωθούν. Βέβαια κάπου αυτά χαθήκανε ε, με τα χρόνια. Ε, το σημαντικό είναι να ξέρουμε τι μπορούμε θετικό να βγάλουμε ε, από αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να τα συνεχίσουμε. Ένα σημείο τώρα όσον αφορά τα, τις στρατιωτικές πτήσεις. Ε, Βεβαίω και για αυτή την περίπτωση εγώ θα πω αυτό που και παλιότερα. Δεν είναι ότι μα λείπουν τα χρήματα, είναι ότι τα χρήματα βρίσκονται σε λάθο χέρια. Ε, το ζήτημα είναι να μοιραστούμε σωστά ε, τα πράγματα. Τώρα, αν πα στον ε, στρατιωτικό και του πει θέλω το δικό σου αέριο χώρο, τον απαιτώ, θα τον δώσει. Αν όμω ε, του πει πολύ ευγενικά, καταλαβαίνει πόσο ανοησία είναι να ακολουθεί τεχλασμένε γραμμέ μία πτήση αντί να πηγαίνει απευθείας από το ένα σημείο στο άλλο και επομένως έλα να καθίσουμε και να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι ε, θα σου πει και αυτός, ναι, ναι, προφανώς, από τη στιγμή που έχουμε κομμάτια του χώρου που δεν χρησιμοποιούνται, οι ώρες που δεν τα χρησιμοποιούμε, γιατί να μην τα μοιραστούμε. και είναι σαφές ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίγουσας ή κατάστασης έτσι κι αλλιώς θα πάρουν πίσω τον εναέριο χώρο, επομένως δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, όσον αφορά την διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ε, λειτουργικών τμήματων εναερίου χώρου, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι να έχουμε εννέα ε, ξεχωριστά φάμπς. Το θέμα είναι να είμαστε σίγουροι ότι τα FABs αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους, συντονίζουν τη δράση τους, αλλά ε, ε, πρέπει και προς τα έξω να έχουν συντονισμό και προς τα μέσα και μεταξύ τους. Ε, βλέπω ότι δεν υπάρχει ακόμα ολοκλήρωση ανάμεσα ε, στο βρετανικό σύστημα και το ε, Ιρλανδικό έστω και αν εσύ το παρουσίασε σαν ένα ενιαίο φαμπ και μέχρι ένα βαθμό κάνουν κάποια πράγματα μαζί. Αλλά όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Τζόρτζ, μπορείς να απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια. <clears throat> αλλά πάντως χαίρομαι για την ωραία συζήτηση που διεξήχθη. Τώρα, για το ε, νέφος ηφαιστιακής τέφρας δεν έχω απολύτως καμία αρμοδιότητα. Προέκυψε το πρόβλημα από την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας στις εναέριες μεταφορές. Αυτό είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΑΣΑ από τη μια μεριά, η Ευρωκοντρόλ και οι άλλοι διεθνείς φορείς αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν μεταξύ των. Τέθηκε το θέμα και στο Μοντρεάλ χθε και σήμερα νομίζω. Ακόμα δεν γνωρίζω ποιε είναι οι αντιδράσει. Γνωρίζω ότι ορισμένοι υπουργοί ήταν δυσαρεστημένοι. Στην ημερησία διάταξη δεν περιλαμβανόταν, αλλά κάποιο σηκώθηκε και είπε ναι, περιλαμβάνεται στα διάφορα. Παρόλο που δεν ήταν επισήμω ε, στην ημερησία διάταξή του, διεξήχθησαν πάντω κάποιε συζητήσει. Θα δούμε ποια πορίσματα προέκυψαν. Πάντως, όπως είπα, το θέμα είναι καθαρά θέμα ασφαλείας. Πώς θα, αντιμετωπίσει, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό ξανά στο μέλλον δεν έχω καμία αρμοδιότητα, όπως είπα. Τώρα, η κατάσταση στην Αμερική, η Λατινική Αμερική, συγγνώμη, είναι σημαντικό σε τραφάμπ. Δεν μπορώ να κινήσω τίποτε. Είναι θέμα περισσότερο των ε, εταιριών και της Κομισιόν, πώς θα διαμορφωθούν δηλαδή οι σχέσεις με τη Λατινική Αμερική το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ολόκληρη Ήπειρο, με την οποία έχουμε στενά πολιτιστικά δεσμά. Αλλά όπως είπα είναι εκτός βελινεκόσμου, μου, μου. Αγαπητή κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Τσικάου, θα είμαι ειλικρινής, αλλά θέλω, πάντα είμαι ειλικρινής, θα το πω όμως όχι διπλωματικά, ας το πω έτσι. Τα ΦΑΜ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις χώρες μέλη δεν πρόκειται να υπάρξουν ευρωπαϊκοί πόροι για τα ΦΑΜ. Έχουν καθήκοντα άσκηση κυριαρχία, όπω έχουν για παράδειγμα αστυνομικά καθήκοντα ε, επί του εδάφου, έχουν και τα καθήκοντα άσκηση του ελέγχου στου εφαίρε, που χρηματοδοτούνται από του φόρου και κυρίω από τα τέλη. Διότι τα αεροπλάνα που πετούν πάνω από την επικράτεια μια χώρα πληρώνουν τέλη και αυτά χρησιμοποιούνται για τον εξυγχρονισμό των δομών ασφαλεία κλπ. Αυτό που είπατε, η κοινοπραξία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτό σημαίνει ότι τότε η κοινότητα ρίχνει λεφτά, αλλά η αγορά software και hardware είναι υπόθεση των χωρών μελών. Δεν είναι θέμα κοινοτική αρμοδιότητας. Υπάρχει ένα μικρό ποσό 20 εκατομμυρίων που θα προσφέρει κάποια βοήθεια, θα προσφέρει κάποιο κίνητρο, αλλά ό,τι και να γίνει, είτε με την ΣΕΖΑ είτε χωρίς, θα χρηματοδοτηθεί από τις χώρες μέλη. Ούτε μπορούν να βγουν και να πούνε ότι δεν θα κάνουμε φαμπ διότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να ενισχυθούν περισσότερο τα φαμπ, αλλά πάντως τα κέντρα ελέγχου οφείλουν να τα χρηματοδοτήσουν οι χώρες μέλη. Για το σκοπό αυτό άλλωστε εισπράττουν τέλη τα πιο δύσκολα θέματα που βλέπω είναι άλλωστε διαφορετικά αναχώρα. Δεν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ένα τυπικό πρόβλημα. Αν θέλω οπωσδήποτε να ψάξω να βρω ένα ε, γενικό πρόβλημα, ένα τυπικό πρόβλημα, θα πω ότι δεν υπάρχουν επαρκή συνεργάτες στο επίπεδο των Υπουργείων για να, τη συνεργασία αυτή. Υπάρχουν χώρες που έχουν τόσο λίγους συνεργάτες στα Υπουργεία, επίσης ε, στις ε, εθνικές αρχές. Για παράδειγμα στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι, έχουν μόνο 70 ε, συνεργάτες στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Εκεί πρέπει οι χώρες μέλη λοιπόν να κάνουν πραγματικά σωστά τη δουλειά τους, να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Παλαιότερα δεν υπήρχαν εθνικές αρχές, υπήρχαν όλα, όλα ήταν μονάχα αρμοδιότητα Υπουργείων. Ε, πρέπει τέλο πάντων οι οργανισμοί και οι φορεί αυτοί να δημιουργηθούν. Και χρειάζεται επομένω να διαθέτουν και χρήματα και συνεργάτε. Ε, κοιτάξτε, είναι όπω είπα αρμοδιότητα και ευθύνη των χωρών μελών. Δεν μπορεί να βγει μια χώρα και να πει δεν μπορώ να κάνω τίποτα διότι δεν έχω κόσμο, δεν έχω προσωπικό. δεν έχουμε λεφτά διότι έχουμε κρίση ε, δημοσιονομική, δεν μπορούμε να βρούμε από τον προϋπολογισμό κτλ. Αυτά δεν μπορούν να ισχύσουν ως ε, δικαιολογίες. Και εσείς ως ευρωβουλευτές θα κληθείτε ε, να συζητήσετε και με τις κυβερνήσεις σας, των χωρών σας δηλαδή, και με τα κοινοβούλια σας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγει μια κυβέρνηση και να πει δεν έχουμε συνεργάτες, δεν έχουμε κόσμο που να ασχοληθεί, άρα δεν μπορούμε να το προωθήσουμε το ΦΑΜ. Τώρα για την Ιορδανία και το Ισραήλ θα σας πω περισσότερα όταν θα τα ξέρω καλύτερα τα πράγματα αυτά. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντως οι τέσσερις χώρες που είναι ε, ήδη ε, χώρες μέλη, δηλαδή Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα, αυτές πρώτα να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν. Έχω την εντύπωση ότι ήδη αυτές οι τέσσερις δεν συμφωνούν. Αλλά ας αρχίσουν τέλο πάντων να συνεργάζονται αυτές οι τέσσερις και μετά βλέπουμε για Ιορδανία και Ισραήλ. Έχω ορισμένες ενδείξεις περί τίνος πρόκειται, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς αυτό. Η μόνη δυνατότητα που έχω εγώ είναι να διαμεσολαβήσω. Να, θα μιλήσω με τους Κυπρίους. Ναι, είχαμε πάει και στην Κύπρο κάποτε. Οι Κύπροι καμιά φορά έχουν και τα δικά τους συμφέροντα τα οποία ε, προσπαθούν με, να προωθήσουν με κάθε τρόπο. Θα πω λοιπόν ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα για τα χρήματα δεν μπορεί να υπάρξει πρόφαση από πλευρά οποιασδήποτε κυβερνήσεως που να πει ότι το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2012 θεωρώ ότι είναι άσχετο, δεν μπορώ να το υλοποιήσω. Το 2012 περιλαμβάνεται στην νομοθεσία και ισχύει και για όποιε χώρε λένε ακόμη ότι κοιτάξτε είναι δύσκολο, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε κτλ. Θα χρειαστεί να συνομιλήσουμε βέβαια με τι ε, κυβερνήσει δεν ε, μπορούμε όμως να δώσουμε να, τη δυνατότητα να υπάρχουν καθυστερήσεις. Συ, Μαριάν, έχεις δίκιο. Τα FAMS είναι ένα στοιχείο, ένα εργαλείο, ένα ενδιάμεσο βήμα προς την ενοποίηση των εθέρων. Το μέγα θέμα είναι, επειδή η Ευρωκοντρόλ είναι απόλυτα άξια να κρατήσει την ασφάλεια αλλά το SS2 είναι παραπάνω από ε, την ασφάλεια και μόνο. Είναι και θέμα, όπως είπα, αύξησης χωρητικότητας, αύξησης αποδοτικότητας, καλύτερης οργάνωσης δηλαδή. Επομένως, οι εθέρες είναι κάτι περισσότερο από ασφάλεια και μόνο. Για τα κέντρα ελέγχου δεν μιλώ για την ώρα ακόμη. Διότι αν αρχίσω να μιλώ για κέντρα ελέγχου, θα ξεσηκωθούν όλοι και θα αρχίσουν να μου λένε ότι θέλεις να καταστρέψεις θέσεις εργασίας. Στη Γερμανία γίνεται τεράστια συζήτηση, λένε να μειωθούν οι ρόλοι των στρατιωτικών, να μειωθεί ο στρατός γενικά. Όλοι η συζήτηση είναι γενικά μείωση του στρατού. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Μόλι πάει να πει κάποιο όμω, Υπουργό Άμυνα, Α, θα κλείσουμε ένα στρατόπεδο, ξεσηκώνονται όλοι τα ομοσπονδιακά κατήρια. Δηλαδή, Α, όχι, όχι σε εμά, όχι σε εμά, να μην κλείσει το στρατόπεδο και θα χαθούν τόσε θέσει εργασία. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια συζήτηση λογική και να δούμε. Τώρα, για το hard και το software. Πρέπει βεβαίω να ενοποιηθούν, αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό δεν θεωρώ επίσης ότι πρέπει να πληρωθεί από του κοινοτικού πόρους, διότι δεν έχουμε τόσα λεφτά. Θα πρέπει να τα κάνουν οι χώρες μέλη μέσω φόρων, μέσω τελών. Κανένας να μην βγει να μου πει ότι δεν έχω λεφτά. Η ιδέα για ακαδημίες κοινή εκπαίδευσης για όλους τους συνεργάτες των κέντρων ελέγχου, αυτό μου φαίνεται σωστό. Ένα άλλο πράγμα είναι η ροή των πληροφοριών, να γίνει πιο αποτελεσματική. Να ε, συμμετέχουν όλοι ταυτόχρονα. Δηλαδή και η εταιρεία και το αεροδρόμιο να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή που ε, σημειώθηκε μια θύελα, για ποιο λόγο καθυστερεί το αεροσκάφος. Να υπάρχει δηλαδή διαρκής ανταλλαγή και ροή πληροφοριών μεταξύ των αεροδρομίων, των εταιριών και καθεξής. Απρόσκοπτη ροή. Βεβαίω αυτό είναι θέμα των τεχνικών. Τώρα, σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλη ιστορία. Υπάρχουν διαφορετικά καθήκοντα που επιβάλλει και η νομοθεσία, είναι διαφορετική και η χώρα. Ο διάδρομος μεταξύ Βοστόνης και Ουάσιγκτον είναι περίπου όσο Παρίσι, Άμστερνταμ, Κολονία, Φραγκφούρτη. Αλλά υπάρχουν τμήματα στην Αριζόνα ή στο Νέο Μεξικό που δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο έλεγχος. Εκεί τους λένε παιδιά πετάξτε όπως θέλετε. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετικές ε, και οι γεωγραφικές συνθήκες. Ο δικός μας έλεγχος μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός, αλλά να πούμε ότι, α, κοιτάξτε, οι Αμερικανοί έχουν λίγους ελεγκτέ, άρα και εμεί χρειαζόμαστε λίγους, αυτό δεν μπορεί να το πει κανεί. Είναι πολύ διαφορετικές συνθήκε εκεί. Εγώ δεν βλέπω ε, κίνδυνο απολύσεω ούτε πιλότων, ούτε εναερίων ελεγκτών. Ίσως ε, σε κάποιες χώρες να είναι λίγοι παραπάνω και σε άλλες χώρες ε, μερικοί παρακάτω από ό,τι χρειάζεται. Μπορούμε να δούμε πώς θα οργανωθούν καλύτερα οι εναέριοι ελεγκτές. Ε, είναι διαφορετικό πάλι το θέμα των σιδηροδρόμων, όπου υπάρχει και το γλωσσικό πρόβλημα. Αλλά εκεί υπάρχει το πρόβλημα το γλωσσικό και, στις, και στους ελέγχους, αλλά όλοι μιλούν αγγλικά τουλάχιστον εκεί. Τώρα, η ανεκτότητα για το περιβάλλον, η φιλικότητα ας πούμε, για το περιβάλλον. Ε, τα πράγματα είναι παρόμοια εδώ, όπως για τα φορτηγά. Μπορούμε να μειώσουμε και να μειώσουμε και να μειώσουμε τους ρήπους, αλλά ε, αγοράζουν ε, όλο και περισσότερα φορτηγά, διότι χρειάζονται όλο και περισσότερα φορτηγά. Είναι μια ατελείωτη ιστορία αυτή. Ναι, όχι, κοιτάξτε μια στιγμή, κύριε Λίχτενμπεργκερ. Εάν καταφέρουμε να κινείται ένα αεροσκάφο από σημείο Α ή σημείο Β ευθέως, χωρίς ζιξάκ, μπορείτε να κάνετε πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις καυσίμων. Εάν οργανώσετε εκ νέου τους εναερίους διαδρόμους, θα δοθεί η σημειο β Ευθέω χωρις ζυξακ μπορειτε να κανετε πολυ μεγαλες εξοικονομησει καυσιμων εαν οργανωσετε εκ νεου τους εναεριου διαδρομους θα δοθει η δυνατοτητα πραγματικα να εξοικονομηθει καυσιμο και επομένω ρήπη. Και αυτό είναι ένα στόχο για όλους μας. Και αυτό ε, θα το θα περιλάβουμε και ξεκάθαρα δεδομένα και στην ε, review που θα κάνουμε. Είναι λοιπόν κάτι επί το οποίο θα εργαστούμε. <clears throat> Θα συζητήσουμε και με τους στρατιωτικούς. Είμαι αντίθετος με οποιαδήποτε έννοια αντιπαράθεσης μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Έχω γνωρίσει βέβαια μερικούς πτεράρχους, λογικοί άνθρωποι μου φαίνονται και πολύ αφοσιωμένοι στο έργο τους. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι όλοι λοιπόν αυτοί οι αξιωματικοί της αεροπορίας θέλουν και καλά να αποκλείσουν ε, ε απολύτως τους χώρους όπου μπορούν να κινούνται μόνο κριτικά αεροσκάφη. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Οτιδήποτε άλλες ερωτήσεις μπορείτε να μου τις στείλετε ηλεκτρονικά. σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά εξαιρετική αυτή η συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Και νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία αποκομίσαμε από την συνάντηση μαζί σου είναι το εξής. Όταν ακούσαμε ότι διορίστηκες ε, στη θέση αυτή, δεν θεωρήσαμε ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ε, αλλά βεβαίως ε, διαπιστώνουμε ότι εσύ, επειδή είσαι εσύ και μπορείς να είσαι τόσο υπομονετικός και τόσο διπλωματικός με τις ε, χώρες, ε, πραγματικά μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Θα είμαστε βέβαιοι ότι θα πιέσει τα κράτη-μέλη όσο πιο πολύ μπορείς και όσο πιο πολύ γίνεται και είμαστε βέβαιοι ότι τελικά θα επιτύχεις. Βεβαίως θα είσαι πάντα εξαιρετικά καλοδεχούμενος οποτεδήποτε είτε εσύ θέλεις να μας πεις κάτι είτε εμείς ε, θεωρήσουμε απαραίτητο να σε ακούσουμε ή να σε ρωτήσουμε κάτι. Σου ευχόμαστε, ε, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σου και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε και θα έχουμε επαφή μαζί σου εις το μέλλον. Okay, colleagues, with you. Εντάξει λοιπόν συνάδελφοι, έχουμε την ε, κυρία Τικάου τώρα. Έχουμε προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα, αλλά εάν η κυρία Τικάου ε, θέλει να μας κάνει αναφορά για την έκθεση της σχετικά με τις εφαρμογές GNSS, παρακαλώ. Και όσοι φεύγετε παρακαλώ να μην θορυβείτε. Κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο που εξετάζουμε είναι η πρώτη ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση για τις εφαρμογές GNSS. Το έγγραφο αυτό δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα. Είναι έγγραφο soft law, όπως λέμε. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Και περιμένουμε και τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το άρθρο 185 της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, θεσπίζει νέες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολιτική διαστήματο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει φυσικά νέες πρωτοβουλίες και να στηρίξει επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, ενώ ταυτόχρονα συντονίζει προσπάθειες για την εξερεύνηση του διαστήματος. Το σχέδιο δράσης GNSS αποτελεί το καρπό μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και καθορίζει ορισμένες προτεραιότητες για την βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης στην ενιαία αγορά. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά μέσα που χρειάζονται για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος. Προβλέπονται επιπρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες ενός δις για μία επιθετία. Οι εφαρμογές του GNSS είναι απαραίτητες για την προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών και μπορούν να έχουν άμεσες συνέπειες σε θέματα μεταφορών, περιβάλλοντος, ασφάλειας μεταφορών, υγείας κτλ. Προτάθηκε και ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Άλλωστε το σύστημα Άγνος λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου του 2009. Πρόκειται για τρεις ε, δορυφόρους και τρεις α, σταθμούς χερσαίους. Το σύστημα αυτό συμπληρώνει το προηγούμενο σύστημα GPS και προσφέρει σημαντικές εφαρμογές και για την ενιαία αγορά αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και οι μεταφορές είναι ένας από τους κλάδους που θα υποφεληθούν σημαντικά από τις εφαρμογές του GNSS. σε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη θέση, την υπολογισμό της ταχύτητας και την συγκέντρωση στοιχείων, αναφορά στοιχείων. Σε αυτούς τους τομείς οι μεταφορές θα υποφεληθούν από τις εφαρμογές GNSS. Και προκειμένου να εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το GNSS, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την έρευνα στον τομέα αυτό. Δυστυχώς, ο προπολογισμό της έρευνας για την ε, σύλληψη και εφαρμογή κάποιων, εφαρμο... κάποιων πρωτοβουλειών, ε, ο προπολογισμό είναι πενιχρός και πολύ σύντομα θα εξαντληθεί. Γι' αυτό και ένα από τα βασικά μας αιτήματα θα πρέπει να είναι συμπλήρωση του προϋπολογισμού. Και όταν μιλούμε για ανακατανομή των ε, μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων στην διάμεση αναθεώρηση, θα πρέπει να ζητήσουμε και συμπληρωματικό ποσό για τη δημιουργία των νέων εφαρμογών. Παρόλο που το πρόγραμμα Γαλιλαίο δεν είναι πλήρως λειτουργικό, προβλέπεται ένα χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2013, που θα περάσει στην ε, λειτουργική φάση με 18 ε, δορυφόρους και αργότερα θα έχουμε 30 λειτουργικούς δορυφόρους. Βέβαια, αν θέλουμε το σύστημά μας να προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες και να διεκδικεί σημαντικό μερίδιο της αγοράς, θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις εφαρμογές. Γι' αυτό και θα πρέπει να ελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές, ιδιωτικές εταιρείε που μέχρι στιγμής αδιαφόρησαν σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Για δύο λόγους κυρίως δεν μπορέσαμε να προσελκύσουμε τους ιδιώτες επενδυτές. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής πλήρης κάλυψη η διαθεσιμότητα και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κονδύλια για την έρευνα είναι πενιχρά. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να συμπληρώσουμε τον προϋπολογισμό, να προσθέσουμε κάποια κονδύλια και ευελπιστώ ότι θα μας υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Άλλωστε, πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια έχουν συνυπογράψει ένα μανιφέστο και πιστεύω ότι για την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό να πολλαπλασιάσουμε τις εφαρμογές του GNSS για να εξασφαλίσουμε σωστή λειτουργία και κατάλληλο μερίδιο αγοράς για το ευρωπαϊκό σύστημα. Ένα άλλο θέμα που αφορά το GNSS είναι ότι ο προπολογισμός έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προβλέπει 25 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θεωρητικά. Για το ICT, επικοινωνία και πληροφορία, έχουμε 3,5 φορές περισσότερα κονδύλια από ό,τι για το GNSS. Παρόλο που το GNSS προσφέρει υπηρεσίες ε, που θα ωφελήσουν περισσότερους τομείς. Έγινε ένας προγραμματισμός για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε τις νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαστήματος και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να πω ότι για τον Ιούνιο περιμένουμε την νομοθετική πρόταση για την ε, πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γκαλιλαίου. Πρόσβαση που θα ρυθμίζεται κρατικά και προβλέπεται και η πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης ε, της Γης, GMES. Αυτά για το 2011. Επίσης για το 2011 προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GNSS και για το ίδιο έτος, το 2011, αναμένεται η πρόταση κανονισμού ε, για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Αυτά ως προς τις νομοθετικές προτάσεις, αλλά έχουν προγραμματιστεί και μη νομοθετικές προτάσεις για το δεύτερο εξάμεινο του 2010. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής θέσης για την εξερεύνηση του διαστήματος. Επίσης, τη μελλοντική ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαστημική πολιτική και η ανακοίνωση Τρίτο μη νομοθετικό έγγραφο είναι η ανακοίνωση που σχολιάζω εγώ στην έκθεσή μου. Το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ε, έχει ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα και την Ινδία, διεκδικώντας όσο το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε επιγόντως της ε, εφαρμογής GNSS, αλλά και επενδύσεις στην ανάπτυξή τους. Επίσης θα πρέπει να περάσουμε στην τελευταία φάση της λειτουργικότητας, λειτουργικής εφαρμογής του προγράμματος Γαλιλαίο. Αλλά για να είναι λειτουργικό το σύστημα, χρειαζόμαστε προηγουμένως εφαρμογές. Και για να έχουμε εφαρμογές θα πρέπει να εφοδιάσουμε περισσότερα κονδύλια τα προγράμματα αυτά. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος για να δημιουργηθούν και εφαρμογέ για τη χρήση του. Ευχαριστώ κύριο Σκούν από το ΕΛΚ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσικάου. Ως εισηγήτρια αναφέρατε πραγματικά όλα όσα απασχολούν τους εισηγητές. Βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό με τους άλλους μεγάλους οικονομικούς ε, παίκτες Κίνα, Ιαπωνία, Ινδίες το ε, GPS χρειάζεται αυτό το σχέδιο δράσης ώστε να οριστούν ξεκάθαρα τα πεδία εφαρμογή. Αυτό είναι σημαντικό και για τις χώρες μέλη ώστε να εξασφαλίσουν και περαιτέρω χρηματοδότηση παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια για το Γαλιλαίο. Είπατε σωστά ότι διατέθηκε ένα δισεκατομμύριο παραπάνω και για μας που ασχολούμαστε με τις μεταφορές, εάν τελικά θέλουμε να είναι λειτουργικό το Γαλιλαίο, έχει σημασία να δούμε πόσο θα βοηθήσει να προωθήσουμε τα FEE συστήματα μεταφορών, για παράδειγμα για προειδοποιήσεις για σημεία εχμής, για μείωση των ρήπων, για ασφάλεια των μεταφορών. Έχουμε τους μεγάλους αυτούς τομείς εφαρμογής. Είναι κρίμα που το Γαλιλαίο το έχει αναλάβει τώρα η Επιτροπή Οικονομικών. Και το μέλλον των συστημάτων διοδίων για τους αυτοκινητοδρόμους θα διασυνδεθεί με τον Γαλιλαίο είναι σημαντικό να υπάρξουν και έλεγχοι για τις επιδοτήσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγχοι ιδιαίτερα για παράδειγμα στον τομέα της γεωργίας. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα εκεί με τα συστήματα πλοηγήσεως ώστε να οριστούν ξεκάθαρα τα πεδία αυτά εφαρμογής. Το ίδιο για την ναυσιπλοεία. Μιλήσαμε μάλιστα σήμερα και μάλλον ψηφίσαμε μάλιστα την ε, ε, έκθεση της κυρίας Μάισνερ για το αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης για τα σκάφη που θα παίξει ρόλο και για την ασφάλεια των σκαφών, ακόμα και οχηματαγωγών και μέσα στα λιμάνια. Έχει λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά ακόμα να γίνει. Ευχαριστώ την κυρία Συγήτρια. Πράγματι θέλουμε να αυξηθούν οι πόροι για την έρευνα. Αλ Καντράουι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ο εισηγητής και ο κύριος, ε, η εισηγήτρια και ο κύριος Κούν είπαν αυτά που στην ουσία θέλω να πω εγώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς σαν Επιτροπή Μεταφορών να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα ε, με το θέμα αυτό. Έστω και αν υπήρξε μια ολίσθηση ας πούμε των, ε, μεταφορών, των αρμοδιοτήτων μεταφορά προς την Επιτροπή. Πρέπει να ασχολούμαστε στο μέλλον και μάλιστα ακόμα περισσότερο. Το σύστημα δυστυχώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ ε, εν μέσω βεβαίως οικονομικής κρίσης. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε. Ξέρουμε ότι το περιθώριο δράσης που έχουμε είναι πολύ περιορισμένο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κυρίως δε ε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις ε, εφαρμογές του Γαλιλαίου ε, στις μεταφορές. Δηλαδή πώς μπορεί ο Γαλιλαίος να μας βοηθήσει έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις μεταφορές και μάλιστα τα στοιχεία αυτά να υπάρχουν όλα σε ένα κείμενο όπως πολύ σωστά μια πρώτη αρχή έχει γίνει στην έκθεση Gross. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μιλήσουμε θετικά. Ε, η κυρία Τικάου επέμεινε ε, σε πολλά σημεία τα οποία συνδέονται με τις μεταφορές και αυτό είναι πολύ θετικό. Ε, την ε, εξωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, ε, την, την αποτελεσματική χρήση των συστημάτων έτσι ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση, να αποφευθούν οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις, οι μεγάλες ουρές κτλ. Πολλά στοιχεία και θετικά, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα. Και θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να αναφερθείτε σε όλα τα στοιχεία του καταλόγου που περιεχόταν στην έκθεση που ανέφερα και εάν ε, έχουν καλυφθεί ή αν πρέπει να προσθέσουμε και κάποια άλλα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τις προτεραιότητές μας. Το σημαντικό είναι να εφαρμοστεί ε, η πρακτικά να εφαρμοστεί επιτόπου δηλαδή αυτός ο κατάλογος. Αλλά δεν θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να μείνουμε μονάχα στα ωραία λόγια ή σε κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι προχωράμε. Ευχαριστώ την εισηγητρία, ευχαριστώ για την παρουσίασή της. Ε, δεν θα επαναλάβω τα όσα ήδη ελέγχθησαν. Ο κ. Χατράου είπε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσον το Γαλιλαίο μπορεί πράγματι να συμβάλλει σημαντικά για την ε, υλοποίηση της Λευκής Βίβλου. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι το Γαλιλαίο θα συμβάλλει σημαντικά. Ε, αυτό που είπε ήδη ο προηγούμενος ο κύριος Κούν ήταν, ε, είναι σωστό, εξεφαστηρίπτου του δηλαδή, που αφαιρέθηκε από τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Μεταφορών το Γαλιλαίο, ειδικά διότι για να ε, προωθηθούν ευφύ συστήματα μεταφορών για την αποφυγή σημείων Στην ε, περιοχή μου ήδη, όχι βέβαια ε, ο Γαλιλαίος δεν υπάρχει ήδη, χρησιμοποιούνται ευφύ συστήματα μεταφορών και ήδη ωφέλει ένα σημαντική. Το ίδιο για την εποπτεία των θαλασσών, ολοκληρωμένη αυτή η πολιτική που ανέφερε πριν ο κ. Κούν είναι επίσης ε, ε, σημαντική και ελπιδοφόρα. Κύριε Λίχτενμπέργκερ, κοιτάξτε, ακούγοντας τα όσα εξήγησε η συγγήτρια, εξακολουθώ να έχω την εντύπωση ότι προφανώς στην ευρωπαϊκή οικονομία η πίστη ότι κάποτε θα λειτουργήσει το Γαλιλαίο και το INSS είναι ακόμα περιορισμένα, η πεποίθηση δηλαδή. Είδε θα, είχαν αρχίσει, θα είχε αρχίσει ήδη η εξέλιξη των εφαρμογών. Δεν γίνεται αυτή η εξέλιξη εφαρμογών. Διότι χρησιμοποιούν ακόμα το παλαιό σύστημα, το GPS, το οποίο το γνωρίζουν όλοι και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για έλλειψη εμπιστοσύνης έλλειψη πεπιθήσεως ότι το πράγμα αυτό θα συνεχιστεί. Αυτό δηλαδή το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό σύστημα ότι πραγματικά θα ανδρωθεί και θα λειτουργήσει. Οι καθυστερήσεις των τελευταίων ετών έδειξαν καθαρά ότι δεν είναι όριμο το σύστημα και δεν οδηγεί επομένω και σε επενδύσεις. Και ούτε θα οδηγήσει εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση των χωρών μελών. Και εδώ εντοπίζεται το κρίσιμο πρόβλημα. Οι χώρες μέλη πολύ απλά δεν έχουν βάλει ακόμα τα πόδια στους βατήρες. Δεν είναι έτοιμες να συνεργαστούν. Ωραία είναι να λέμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι, αλλά πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Διακινδυνεύουμε να δούμε να, είναι, να εμφανίζεται εν τέλει ένα θνησιγενές σύστημα. Εάν δεν εμπλέκεται η ιδιωτική οικονομία, μένουν όλα αυτά στη θεωρία. Και είναι όλα κούφια λόγια. Είμαι υποχρεωμένη να τα πω έτσι ξεκάθαρα, διότι εγώ ενδιαφέρομαι πράγματι να λειτουργήσει εν τέλει το σύστημα. Πώς όμως θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων εφόσον δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Αυτά τα λένε και στις χώρες μέλη, αυτά τα λέει και τα σκέφτεται και η οικονομία, η ιδιωτική οικονομία. Εκεί βρίσκω το, ότι είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα ήταν κάποιος. Μπορεί να μα απογοητεύει η απουσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Σίλβια, θέλει να απαντήσει ε, στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις στα σχόλιά τους και τις ε, προτάσεις τους. Αυτή είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η έκθεση θα εκπονηθεί σύντομα και ήδη είχα αρκετές ε, συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, και ε, από όσο καταλαβαίνω θα στηρίξουν την προσπάθειά μας να ζητήσουμε επιπρόσθετο συμπληρωματικό προϋπολογισμό θα στηρίξουν τις κοινέ ε, πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναμειχθεί αποτελεσματικότερα και ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να εξευρεθεί ο κατάλληλος μηχανισμός έτσι ώστε να διασφαλιστούν ε, τα ε, απαραίτητα εχέγγυα προς τους επενδυτές και ότι η όποια θετική επένδυση κάποια στιγμή στο μέλλον ε, θα επιβραβευθεί από την αποτελεσματική χρήση του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει αρκετές ε, επιλογές ε, για την ανάπτυξη του συστήματος θα, υπάρξουν, θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός δράσεων ε, τις ε, οποίες ε, θα επικεντρώσουμε στην προσπάθειά μας για καλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα με όσο γίνεται μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας και όσο γίνεται μεγαλύτερη βελτίωση του τομέα των μεταφορών. Το σύστημα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κοινού με την στρατηγική του ενιαίου ε, ε, ουρανού ε, και την ΣΕΖΑΡ, θέματα τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Στον τομέα των μεταφορών υπάρχουν αρκετές δράσεις οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη του συστήματος αυτού. Από την άλλη πλευρά, θα αναλύσω με τον κατάλογο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως θα έχουμε και τις δικές μας προτάσεις Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή Μεταφορών θα οργανώσει γύρω στα τέλη του τρέχοντος έτους μια ακρόαση όσον αφορά την ανανέωση του συστήματος Γαλιλαίου και τις εφαρμογές του συστήματος GNSS. Και νομίζω ότι θα είναι κεφαλαιόδου σημασίας ε, να έρθει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και με έναν, μια πρόταση κανονισμού ε, όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες μέσω αυτού του συστήματος και βεβαίως πολλές από τις ευρωμογές θα συνδέονται με τις μεταφορές. Για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Ε, περιμένω και περαιτέρω σχόλια και προτάσεις και παρατηρήσεις. Ελπίζω ότι θα έχετε ενδιαφέρουσες τροπολογίες αργότερα. Και τέλος, πιστεύω ότι χρειάζεται πραγματικά η Ευρώπη το σύστημα Γαλιλαίος έτσι ώστε να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε αποτελεσματικά συστήματα. Άρα θα πρέπει να στηρίξουμε και τη βιομηχανία η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί, να συμμετέχει ενεργά ε, στις διαδικασίες αυτές. Θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ε, να δοθούν κίνητρα στην βιομηχανία έτσι ώστε ε, να αρχίσει να ασχολείται με το θέμα και βεβαίως να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τον τρόπο να κινητοποιήσουμε την κριτική μάζα των χρηστών που θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τικάου. Θα περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις πρωινές μας εργασίες. Τρεις το απόγευμα θα σας βρω. Ε, Τζούλιετ, εσύ θα παίξεις σε πρωταγωνιστικό ε, ρόλο πάλι. Τρεις το απόγευμα.